Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε παρά το μικρό αριθμό των ευρωβουλευτών. Όπως ξέρετε η συνεδρίαση αναμεταδίδεται διαδικτυακά. Σήμερα προβλέπονται δύο ακόμη πάνελ το πρώτο αφιερώνεται στο θέμα της ασφάλειας των τεχνολογιών πληροφορικής των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και το δεύτερο τμήμα της δημόσιας ακρόασης στον ρόλο της κοινοβουλευτικής εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών μετά τις καταγγελίες για τις μαζικές παρακολουθήσεις. Αυτά, αυτό προβλέπει το πρόγραμμα της Δημόσιας Ακρόσης και δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Παρακαλώ να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και να ξεκινήσουμε. Έχουμε εδώ τέσσερις εμπειρογνώμονες. Θα ακούσουμε τις παρουσιάσεις του κυρίου Ρόλτ Πρινς, που είναι διευθυντής και συνειδητής της Fox IT, μιας εταιρείας που εντοπίζει από, ε, προλαμβάνει ή αποτρέπει ε, παραβιάσεις και παγιδεύσεις ε, των συστημάτων ε, στα κοινωτικά θεσμικά όργανα. Είχαμε και την περίπτωση της Belgacom. Έχουμε τον κύριο Φρέντι Ντεζέρ που είναι επικεφαλής της ομάδας αντιμετώπισης διοργανικών έκτακτων περιστατικών σε θέματα πληροφορικής, ΣΕΡΤ ε, υπεύθυνο για την ασφάλεια των, των συστημάτων πληροφορικής ε, των θεσμικών οργάνων ε, με αποστολή την πρόληψη, εντοπισμό, αντικατάσταση, αντίδραση και διόρθωση δόλων και κακόβουλων επιθέσεων που πλήττουν την ακερότητα των συστημάτων. Επίσης έχουμε τον κύριο Βιλέλα που είναι Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού της Διεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια και για τις πληροφορίες, επικοινωνίες και πληροφορίες και τον κύριο Βιλέλα που είναι αξιωματούχος ασφάλειας της EU LISA που διαχειρίζεται τα συστήματα VISIS και Eurodac με πολλά ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία που θα πρέπει να εξασφαλίζονται, να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία τους. Θα δώσω το λόγο για ένα δεκάλεπτο στον κάθε εμπειρογνώμονα, μετά θα έχουμε ένα γύρο ερωταπαντήσεων και συζήτησης και θα μπορέσουμε να καλύψουμε και πολλά άλλα θέματα. Κύριε Πριντς, παρακαλώ, είστε ο πρώτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πράγματι. Έχω προετοιμαστεί για τη συζήτηση μαζί σας. Πράγματι, Ερευνήσαμε την Belgacom και το σχετικό περιστατικό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αντιλαμβάνεστε πως ε, είναι θέμα του πελάτη να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες. Έχω κάποιες γενικές παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Έχουμε εμπλακεί κάποιες φορές σε έρευνα περιπτώσεων κατασκοπίας και αυτό το οποίο βλέπουμε, ε, αν το αναλύσουμε στο τι μπορούν να κάνουν οι πελάτες όσον αφορά την πρόληψη, ανείχνευση και αντίδραση, ε, έχουμε σημαίνει κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας. Π.χ. αντίδραση είναι η δικιά μας ε, δουλειά. Αν σε έναν οργανισμό θεωρούν πως υπάρχει κάτι ύποπτο και θέλουν να καταλάβουν τι γίνεται, Έχουμε τεχνολογία DPI που ψάχνει το τι γίνεται και μετά ξεκινάει μια αρκετά πολυδάπανη έρευνα. Χρειάζεται πάρα πολλούς πόρους για να δούμε το τι συμβαίνει και τι συμβαίνει συνήθως. Κατά κανόνα ο πελάτης ε, έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον δικό του πελάτη ή το κράτος το οποίο χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του. Δηλαδή συνήθως θέλει να καθαρίσει το δίκτυό τους και αυτό κάνουμε, αλλά βλέπετε πως υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν γιατί δεν υπάρχει άμεση πρόθεση έρευνας. Οπότε Πολλές φορές η έρευνά μας ε, τελειώνει με περισσότερες ερωτήσεις όπως ποιος το έκανε, τι πληροφορίες πήρε και τι στόχο είχαν. Αν το δείτε κάπως ε, ευρύτερα είναι κρίμα να μπορούμε να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις. Μετά έχουμε και το θέμα της ανείχνευσης Πολλοί οργανισμοί προσπαθούν να βρουν το τι συμβαίνει στο δίκτυό τους. Όπως ξέρετε ε, μπορούν να προσληθούν οι υπολογιστοί και πρέπει να υπάρξει ένα περιβάλλον εντοπισμού και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πως υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που αναφέρθηκαν και στον τύπο που μάλλον είχαν κάποιο κακόβουλο λογισμικό, αλλά κάνουν μόνοι τους την έρευνα και μετά λένε το τσεκάραμε και δεν υπάρχει τίποτα και δεν τρέχει τίποτα, ηρεμήστε. Κάπως περίεργο, γιατί αφενός έχουμε οργανισμούς, υπηρεσίες ασφαλείας που ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό, πολύ εστιασμένο, εστιασμένο στο να μην ανοιχνεύεται, και κάποιοι άλλοι αγόρασαν ένα κουτί το οποίο κουτί δεν βλέπει τίποτα οπότε λένε αυτοί είμαστε εντάξει και με, με οργανισμούς που δεν ξέρουν τίποτα για τα συγκεκριμένα γεγονότα, δεν έχουν τεχνικούς δείκτες προσβολής ε, του δικτύου και βγάζουν κάποιες ανακοινώσεις ε, τύπου και λένε πως είναι σίγουροι πως δεν έχουν πληγή. Ε, αν είναι το σίγουροι βεβαίως εμείς θα τους προσλαμβάναμε. Και μετά υπάρχει η φάση της ε, πρόληψης ε, που είναι επίσης ενδιαφέρουσα. Έχουμε πολλούς πελάτες ε, που προσπαθούν να είναι ασφαλείς και έχουμε ειδικό εξοπλισμό, ειδικά εκεί όπου είναι κρίσιμο το θέμα της ασφαλείας, π.χ. στα δίκτυα της ενέργειας. Εξάγουμε πολλά τέτοια πράγματα σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι στην Ευρώπη. Και δεν είναι ότι δεν προσπαθούμε αλλά φαίνεται πως είμαστε αφελείς και δεν ε, σκεφτόμαστε πως ε, θα υπάρξει τέτοια επίθεση στην Ευρώπη. Επίσης βλέπουμε πως ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που είναι, διαθέσιμ, που είναι διατεθειμένα να επενδύσουν έχουν ένα πρόβλημα με την πρόσληψη προσωπικού και αγοράς υλικού. Ένας λόγος μπορεί να είναι πως το σύστημα ευρωπαϊκών διαγωνισμών ε, δεν βοηθάει γιατί καταλήγουν ε, στον μειοδότη, κάτι το οποίο δεν σημαίνει πως είναι η καλύτερη λύση. Και επίσης ε, βεβαίως υπάρχει και ένα ζήτημα... Έχουμε κάνει μια μελέτη σκοπιμότητας για εξοπλισμό κρυπτογράφησης εξοπλισμό κρυπτογράφηση σε ολόκληρη την αλυσίδα όταν χρειάζεται να προστατευτούν κρατικά μυστικά. Και βεβαίω έχουμε και ένα κατάλογο εγκεκριμένων προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντό της ευρωπαϊκή Ένωσης για τους χαρακτηρισμούς ε, απόρριτο, άκρο απόρριτο, εμπιστευτικό. Τα πράγματα τα οποία βεβαίως ε, κοστίζουν ε, για τηλέφωνα μιλάω τώρα επίσης, τα οποία όμως δεν ξέρω εάν α, αξίζει τον, κόσμο να τα, τον κόπο να τα αγοράσετε εσείς ως ε, βουλευτές, είναι και πάρα πολύ ακριβά, αλλά είναι πάρα πολύ ασφαλή. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θέλει κανείς να επενδύσει για να αποτρέψει την ε, κατασκοπία. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τεζέρτο, το πολύ για 10 λεπτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομα εισαγωγή για το ΣΕΡ, την ομάδα αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην πληροφορική, ποια είναι τα καθήκοντά μα ε, και οι αρμοδιότητέ μα. Είναι διοργανική η ομάδα κρούσης ε, του ΣΕΡΤ και στόχο έχει να βοηθήσει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να αντιμετωπίσουν ε, απειλές στον κυβερνοχώρο. Είναι μια ολιγομελής ομάδα, 15 μελής, με εμπειρογνώμονες που συστήθηκε πριν από μια διετία και μάλιστα εμπίπτει στη Γενική Διεύθυνση ε, Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην κατευθυντική ομάδα τη διοργανική. Μεταξύ των πελατών μας εντάσσονται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΝΙΣΑ, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, και άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Και φυσικά προσπαθούμε να ε, κρατήσουμε τη λειτουργικότητα των ε, δικτύων τους ε, και την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Επίσης, προσφέρουμε βοήθεια στον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων και στην άμεση αντιμετώπιση τους. Σε διοργανικό και διεθνές επίπεδο ε, συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους δυνατούς εταίρους και εξασφαλίζουμε και ένα συντονισμό μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και αυτή είναι η προστιθέμενη αξία μας. Έχουμε λοιπόν στενή συνεργασία με τους ε, εμπειρογνώμονες ασφάλειες ε, κάθε θεσμικού οργάνου και έτσι προσπαθούμε να διεκπαιρεώσουμε την αποστολή μας. Βέβαια, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα είναι πολύ σημαντική στόχοι γιατί μπορούν από αυτά τα όργανα να κλαπούν οικονομικές, πολιτικές πληροφορίες, να εκδηλωθεί ακτιβισμός, πολιτική δυσαρέσκεια. Αυτό είναι βέβαια το ίσονο σημασίας πρόβλημα, αλλά είναι σίγουρα στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων. Έχουμε τρία είδη υπηρεσιών. Καταρχήν ε, προληπτικού χαρακτήρα, βοηθούμε τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να αποφύγουν στο μέλλον προβλήματα, να εντοπίσουν ποια είναι τα επικίνδυνα λογισμικά. Επίσης, αντλούμε διδάγματα από τις εμπειρίες άλλων κοινοτικών θεσμικών οργάνων, ώστε να βρούμε μηχανισμούς προστασίας. Ό,τι αφορά τον εντοπισμό, συγκεντρώνουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές, είτε από τα ίδια τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, όταν υφίστανται επιθέσεις και έχουμε σχετισμό και με άλλα κοινοτικά όργανα. Λαμβάνουμε από τα εθνικά σέντρα, τις εθνικές ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, με πολύ καλή συνεργασία μαζί τους και επίσης από, από τον ίδιο τον κλάδο για την ασφάλεια των ε, τεχνολογιών πληροφορικής. Επίσης έχουμε και στατιστικά στοιχεία. 650 ε, κρούσματα είχαμε ε, κόδωνες κινδύνου, είτε για διάφορα κακόβουλα λογισμικά, για κλοπή διαπιστευτηρίων. Γενικώ είναι ευάλωτα τα συστήματα και με τα στατιστικά που συγκεντρώνουμε βοηθούμε τα θεσμικά όργανα να αντιδράσουν στα έκτακτα περιστατικά. Ε, βέβαια και τα κοινωτικά όργανα μπορούν να εντοπίσουν τέτοια κρούσματα και να μας ενημερώσουν ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις κυβερνοεπιθέσεις. Όταν έχουμε ένα σοβαρό κρούσμα, ένα σοβαρό συμβάν και παραβίαση συστήματος, μπορεί οποιοδήποτε θεσμικό όργανο να μας καλέσει ε, να βοηθήσουμε. Τότε συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες από τα πιο όρημα θεσμικά όργανα και ε, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε εμπειρογνώμονες από τα πιο μεγάλα θεσμικά όργανα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Επίσης έχουμε επαφές με το Εθνικό Δίκτυο ε, Προστασίας των Δικτύων. Πέρυσι είχαμε τέτοιες 10 υποθέσεις ε, όπου η ομάδα μας στο ΣΕΡΤ χρειάστηκε να εξασφαλίσει κάποιο συντονισμό σε περίπτωση που είχαμε σοβαρά προβλήματα. Εν κατακλείδη να πω ότι η ομάδα μας ΣΕΡΤ είναι μια νεοπαγής ε, ομάδα κρούσης ε, που προσπαθεί να επιφέρει μια προστιθέμενη αξία στη δράση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και έχουμε ε, ένα εμπεδομένο σύστημα και συντονισμένο συγκέντρωση πληροφοριών από τους καλύτερους εταίρους που μπορούμε να βρούμε στον κλάδο. Και αυτό που είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτή η 15 μελής ομάδα που θα μεγαλώσει στο εγγύς μέλλον είναι προσιλωμένο στην ε, ασφάλεια και στην αναβάθμιση της ε, προστασίας και της ασφάλειας των κοινωτικών θεσμικών οργάνων έναντι επιθέσεων στον χώρο. Ευχαριστώ κύριε Δεζέρε. Ο τρίτος μας ομιλητής είναι ο κύριος Βιλέλα, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ΆΙΤΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ε, μιλήσω στα γαλλικά και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους της Ιταλικής ε, Δερμηνίας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι ο τρίτος ε, στη σειρά μετά από τον εισηγητή του ΣΕΡΤ, του Κέντρου Επίγουσες, μάλλον Αντιμετώπισης Επιγόντων Αναγκών στην Πληροφορική, διότι το σύστημά μας βασίζεται στις δράσεις του σε αυτό το τομέα, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, βασίζεται στην διοργανική συνεργασία. Να πρόκειται για ένα θεμελιώδες στοιχείο για μας. Από τον Απρίλιο το Κοινοβούλιο προεδρεύει της Διοργανικής Επιτροπής για την Πληροφορική και στο πλαίσιο αυτό το Κοινοβούλιο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για κοινέ ενέργειε που ξεπερνούν κάπως την συνεργασία που είναι σημαντική και θεμελιώδης στο εσωτερικό του ΣΕΡΤΕ. Το Κοινοβούλιο πρότεινε να γίνουν προσπάθειες για την ανέβρεση λύσεων που να είναι κοινέ. Δηλαδή να υποδομήσουμε κάποιες δομές κοινές ώστε να προστατευτούν καλύτερα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτές οι προτάσεις η Γενική Διεύθυνση ΤΕΚ τις υπέβαλε στη Διοργανική Επιτροπή και επί τη βάση ψηφισμάτων που έχει υιοθετήσει το Ευρωκοινοβούλιο το περασμένο Ιούλιο, οπότε και υιοθέτησε δύο ψηφίσματα όσον αφορά την ασφάλεια στην πληροφορική, την κυβερνοασφάλεια, προτείνοντας μια πιο ισχυρή συνεργασία ανάμεσα στα όργανα, αλλά και μέσα στα ίδια ψηφίσματα περιλαμβάνεται η ιδέα ε, μιας, ενός ε, νέφους, κοινού νέφους. Η Γενική Διεύθυνση ΤΕΚ, συμμερίζεται αυτή την πρόταση του Κοινοβουλίου και γι' αυτό και επισήμως ε, τύπης υπέβαλε αυτήν την ε, πρόταση στο πλαίσιο των διαφορών επιτροπών, ε, αρμοδίων επιτροπών. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ως πρόεδρος της Διοργανικής Επιτροπής για την Πληροφορική, σε αυτό το ρόλο μου, περιμένω με ανυπομονησία τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στο του Inquiry διότι πιστεύω πως όλες οι ενδείξεις που θα περιλαμβάνονται στο ψήφισμα και στην έκθεση ε, που θα εκπονηθεί στο τέλος αυτών των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της Διοργανικής Επιτροπής για την Πληροφορική. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο σχέδιο για την ασφάλεια της πληροφορικής μέσα στο εντός μάλλον του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό που μπορώ να πω και όπως εξάλλου ήδη το είπε ο συνάδελφος του ΣΕΡΤ, κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ασφάλεια στην πληροφορική. Αυτό είναι προφανές. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ITEC στο Κοινοβούλιο έχει ένα επίπεδο παρέμβασης που αντιστοιχεί στα διεθνή πρότυπα και κριτήρια. Ότι δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς είναι ενέργειες που αντιστοιχούν σε πρότυπα διεθνή. Ε, επίσης θα πρέπει να πω, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι περήφανος γι' αυτό. Θα πρέπει να πω ότι καταφέραμε να αντικρούσουμε κάποιες επιθέσεις στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Αλλά πέρα από αυτό θα έλεγα ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι όσον αφορά τα πρότυπα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο, όπως ξέρει και ο κύριος Ντεσέρ, το Κοινοβούλιο συνεργάζεται πολύ με το ΣΕΡΤ. Φυσικά ε, ο τομέας αυτός αποτελεί διαρκή πρόκληση και γι' αυτό και συμμετέχουμε διαρκώς σε σεμινάρια για την ανανέωση των γνώσεων ε, στον τομέα. Και όντως η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής ε, είναι σε θέση να κατανοήσει ποια είναι τα προβλήματα ασφάλειας τι είδους επιθέσεις μπορεί να υποστούμε ή αν είμαστε υπό επίθεση να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Ακόμα και αν κάποιες φορές όλες αυτές οι ενέργειες καθίστανται ε, δύσκολες λόγω ή χάρη στους κανόνες της προστασίας των δεδομένων. Δεν μπορούμε δηλαδή να παρέμβουμε τελείως ελεύθερα. Τέλος, η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΙΤΕΚ e e τα τελευταία δύο χρόνια πρότεινε δύο πράγματα εντός του Κοινοβουλίου και ε, προς αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα και ενεργούμε. Από τη μια πλευρά να γίνει μια αναθεώρηση των κανόνων που υπάρχουν στον τομέα και από την άλλη και κυρίως ίσως να υιοθετηθούν νέοι κανόνες που θα καλύψουν τα κενά. Διότι για να γίνει σωστή και νόμιμη δράση στον τομέα της ε, ασφάλειας της πληροφορικής, ε, εγώ θέλω πάντοτε μια νομική βάση που μας επιτρέπει παρεμβάσεις τέτοιου τύπου. Η δεύτερη πρόταση όπως γνωρίζουν οι πολύ καλά οι ευρωβουλευτές η ένταξη της ασφάλειας της πληροφορικής στο πλαίσιο μιας γενικότερης σφαιρικής πολιτικής ασφαλείας. Γιατί θεωρούμε στην ΓΑΜΑ ότι η ασφάλεια της πληροφορικής δεν μπορεί να είναι ξεχωριστή από μια γενικότερη αντίληψη για την ασφάλεια. Και αυτό θα πρέπει να γίνει. Κατά τα λοιπά, η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ είναι σε θέση να υλοποιήσει διάφορες ενέργειες και προγράμματα αυτόνομα, αλλά όπως όλες οι μεγάλες διοικητικές δομές του κόσμου δεν είμαστε σε θέση εμείς να δημιουργήσουμε υποδομές πληροφορικής και όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με ειδικευμένε εταιρείε στον τομέα της τεχνολογίας επί τη βάση βεβαίως του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτές είναι οι βασικές γραμμές λοιπόν της ε, δράσης της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ e Φυσικά είμαι έτοιμος να απαντήσω σε πιο λεπτομερείς ερωτήσεις εάν είναι απαραίτητο. Για να κλείσω κυρία Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, επιμένω στο εξή σημείο. Το ίδιο όπως στην αρχή της ομιλίας μου ότι η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ βασίζεται κυρίως και θα ήθελε να ενισχύσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη συνεργασία τη διοργανική. Yes, thank you, Mr. Villela. I note that you have taken the ultimate... Βλέπω πως έχετε λάβει το απόλυτο μέτρο ασφαλείας για τις σημειώσεις σας. Είναι χειρόγραφες. Μάλιστα ερχόμαστε στον κύριο Ζαπαλιώνε, ο οποίος ε, εργάζεται στην υπηρεσία Λίζα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Έχω και μια παρουσίαση κάπου. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, λέει η πρόεδρος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Λούκα Τζαμπαλιώνε. Ασχολούμαι την Δουλεύω στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογικών Πληροφοριών Μεγάλης Κλίμακας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι μας ζητήσατε να αναφερθούμε στο ζήτημα της ασφάλειας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τώρα δεν θα αναφερθώ στο τι κάνει η υπηρεσία μου μακρόν. Μια σύντομη εισαγωγή θα κάνω. Μετά το πληροφοριακό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούμε, το ζήτημα, το περιβάλλον ασφαλείας και τα τρία συστήματα τα μεγάλα πληροφορικής και μετά κάποιες συστάσεις για το πώς θα μπορέσουν να βελτιώσουν την πληροφοριακή ασφάλεια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Ελίζα συστάθηκε με τον κανονισμό 1077 του 2011 και είναι η διαχειριστική αρχή πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης ε, κλίμακας στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών, δηλαδή το σύστημα Schengen 2, το Eurodac, το Συνοδεκτικό των και το σύστημα Visa. Είμαστε υπεύθυνοι για την ε, επιχειρησιακή διαχείριση και την ασφάλεια των κεντρικών συστημάτων και για το σύστημα επικοινωνίας, το οποίο συνδέει τα κεντρικά συστήματα με τα κατατόπους. Για να σας δώσω τώρα κάποια νούμερα. Το σύστημα πληροφοριών Schengen 2 συνδέεται με 30 κράτη-μέλη της Schengen και τη Eurojust και τη Europol και πάρα πολλά εθνικά δίκτυα Επιβολή του νόμου. Το σύστημα βίζας συνδέεται με 29 κράτη-μέλη, κυρίως με, το Υπουργείο, με τα Υπουργεία Εξωτερικών και βρίσκεται και σε αρκετές περιοχές του κόσμου, όπως την Αφρική και τη Μέση Ανατολή και προσεχώς και στην Νότια Αμερική και τη Ρωσία. Το Ευρωπαϊκό Δακτυλοσκοπικό Σύστημα για το Άσλο καλύπτει 32 χώρες και αφορά κυρίως ζητήματα μετανάστευσης. Βλέπετε λοιπόν πως υπάρχει μία διασύνδεση με τα εθνικά συστήματα και κάποια περιφερειακά επίσης. Επίσης ανέφερα και το δίκτυο επικοινωνιών που δεν είναι σύστημα, είναι ένας δέκτης ασφαλούς ε, μεταφοράς δεδομένων θα έλεγα πως είναι το ελάχιστο και είναι ένα καλώδιο το οποίο δεν ε, παρέχει ασφαλή σύνδεση. Το μοντέλο ασφαλείας βασίζεται σε μια απλή ιεραρχία. Υπάρχουν κανονισμοί του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, κανονισμοί ασφαλείας και βεβαίως εποπτεύεται και προβλέπεται και για εμάς και για κάθε πληροφοριακό σύστημα ποιες είναι οι προδιαγραφές ασφαλείας οι οποίες πρέπει να πληρώνει κάθε σύστημα. Η νομική βάση λοιπόν είναι αυτή η οποία μας δίνει τις κατευθύνσεις για το πώς θα έχουμε ασφάλεια. Η ιεραρχία είναι φτιάχνουμε σχέδια ασφαλείας και αναπτύσσουμε κάποιες διαδικασίες και πολιτικές ασφαλείας για να έχουμε ε, ιεραρχικά ε, κάποιες διαδικασίες. Επίσης η Λίζα αναπτύσσει ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου γιατί βεβαίως οι απαιτήσει που προκύπτουν από την νομοθεσία δεν μπορεί να είναι οι μόνε απαιτήσει. Όπω ανέφερε και ο συνάδελφο από την Γενική Διεθνή έχουμε και κάποιε προδιαγραφέ ασφαλεία για να έχουμε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για το πώ θα εφαρμοστεί τεχνικά η ε, ασφαλεία. Το μοντέλο ασφαλείας λοιπόν από μια πιο τεχνική σκοπιά προβλέπει κάποιες βασικές αρχές που λειτουργούν. Τα τρία κεντρικά συστήματα έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην συνδέονται με το διαδίκτυο, αλλά μόνο με εξοδοτημένα θεσμικά δίκτυα μέσω κάποιων ελεγχόμενων εθνικών διαπαφών. Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την διασύνδεση με τα κράτη-μέλη, μέσα στο κράτος μέλος, αυτό το οποίο ορίζουμε δηλαδή το όριο. Είμαστε λοιπόν υπεύθυνοι ε, για την ασφάλεια από τα κεντρικά συστήματα μέχρι τη σύνδεση με τα κράτη-μέλη. Από το όριο αυτό περιέγραψα και μετά είναι πλήρως υπεύθυνα τα κράτη-μέλη για την ασφάλεια των εθνικών τους δικτύων. Ενώ τα τρία ε, συστήματα μεγάλης κλίμακας παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Όπως βλέπετε από τα τρία βασικά σημεία που έχω υπογραμμίσει έχουμε μια εφαρμογή των όσων προβλέπονται από πρακτικές ασφαλείας και διεθνείς προδιαγραφές. Παρά το ότι όπως είπα δεν προβλέπονται στην νομική βάση. Τώρα περνάμε στην τελευταία διαφάνεια με κάποια μέτρα ασφαλείας τα οποία κατά την άποψή μας μπορούν να συνεισφέρουν στην βελτίωση του καθεστώτος Φελίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Τέσσερις ε, βασικοί τομείς ε, βελτίωσης ε, υπάρχουν. Ο πρώτος είναι να καθορίσουμε προδιαγραφές ασφάλειας πληροφορικής ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο για μια προσέγγιση σε όλο το μήκος του δικτύου. Αυτό το άκουσα και ε, από τον κύριο εδώ πέρα δίπλα μου. Ε, αυτό το απάκρισάκι άκρη θα τα ακούτε συνεχώς. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας τεχνικός φορέας ο οποίος θα παρακολουθεί και θα εφαρμόζει αυτές τις προδιαγραφές και θα συμπεριλαμβάνει και τα θεσμικά όργανα και τις εθνικές αρχές για να εγγυηθούμε ένα ομοιογενές αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας. Δηλαδή, για να έχουμε ασφάλεια από τα κεντρικά συστήματα όπου βρίσκονται οι βάσεις δεδομένων μέχρι τον τελικό χρήστη που καταναλώνει τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα κεντρικά συστήματα. Η δεύτερη σύσταση είναι να αναπτυχθεί μια τυποποιημένη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου για να διασφαλίσουμε πώς θα εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας ιδιωτικής ζωής για να υπάρξει μια κατανομή του προϋπολογισμού και των πόρων. Εν ολίγης, να βρούμε τα σωστά αντίμετρα τα οποία θα είναι και προσιτά από πλευράς κόστους. Πρέπει να προστατεύονται οι πληροφορίες βεβαίως με κάποια μέτρα ασφαλείας, αλλά πρέπει να βρούμε τα σωστά και αυτό θα γίνει μέσω μιας αξιολόγησης κινδύνου. Έτσι μπορούμε να επιτύχουμε την γνωστή ε, αρχή ασφάλεια από τον σχεδιασμό. Τρίτη σύσταση είναι να προβλεφθεί στον κύκλο ζωής των συστημάτων πληροφορικής μια διαδικασία πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης ασφάλειας. Όπως κάνουμε, παραδείγματος χάρη, με τα αυτοκίνητα τα οποία περνάνε εκταίο, επανειλημμένα, όταν τα συστήματα πληροφορικής ε, γίνονται πιο παλιά, είναι πιο ευάλωτα σε νέες απειλές, ειδικά όταν το επίπεδο απειλής είναι υψηλό, όπως παραδείγματος χάρη όταν είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Τέλος, τελευταία σύσταση. Είναι να δούμε ε, τις έννοιες της διαχείρισης ε, ταυτοποίησης ε, και ένα μηχανισμό ισχυρό όσον αφορά την ταυτοποίηση των πληροφοριών για να είμαστε σίγουροι πως οι πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες ανα πάσα στιγμή από οποιονδήποτε πρέπει να έχει πρόσβαση και όχι σε ε, Και εδώ πέρα σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζαμπαλιώνε. Περάμε τώρα στο γύρο των ερωτήσεων και της συζήτησης. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση προς τους ε, καλεσμένους μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο της Προέδρου. I mean, the NSA has no limits, Φαίνεται ότι δεν ε, γνωρίζει όρια η NSA. Θα ήθελα να επισημάνω ότι διενεργούμε έρευνα μετά από ισχυρισμούς για μαζική παρακολούθηση, κατασκοπία, υποκλοπές, παρακολουθήσεις ε, τηλεφωνικών συνομιλιών και είχαμε ειδική ε, συνεδρίαση για την Belgacom που μάλιστα επηρέαζε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί τα προγράμματα και εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε είναι από τη Microsoft, την Apple και είχαμε καλέσει και προσώπους ε, των εταιριών αυτών σε προηγούμενες συνεδρίες. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω και να λάβω απαντήσεις για το τι συμβαίνει εδώ, πόσο εμείς έχουμε επηρεαστεί από τέτοιες ε, παραβιάσεις. Αν έχετε εντοπίσει τέτοιες παρεμβολές και αν όχι, γιατί δεν τα καταφέρατε. Τέτοιου πληροφορίες θέλουμε να ακούσουμε εδώ. Γιατί εσείς επικεντρωθήκατε περισσότερο στα μέτρα πώληση. Ωραία αυτά, αλλά φαίνεται ότι δεν λειτουργήσαν, γιατί οι δυνάμει εντό εισαγωγικών ε, είναι πολύ ισχυρότερε ε, οι εξωτερικέ δυνάμει. Τέτοιε απαντήσει λοιπόν δεν έχω λάβει μέχρι στιγμή. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Κλοντ Μωράε. Ξέρετε ότι δύο λεπτά προβλέπετε για τον κάθε ομιλητή, δύο λεπτά προβλέπονται, αυστηρά δύο λεπτά. Το ίδιο δίλεπτο ισχύει και για τους καλεσμένους για τις απαντήσεις τους. Θα έχουμε ένα γύρο λοιπόν με τον εισηγητή και τους και και κατόπιν με τους ε, λοιπούς ευρωβουλευτές αν απομείνει χρόνος για δεύτερο γύρο. Και θα επιτρέψω για συγκεκριμένα θέματα και συμπληρωματικές ερωτήσεις αν χρειαστεί. Ο Κλοντ Μωράης. Πάντως ε, και εγώ θα ήθελα όπως είπατε, να απαντηθούν αυτές οι απορίες μας. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό που ερευνούμε στην περίπτωση αυτή είναι τι συνέβη σε σχέση ε, του ισχυρισμού, όχι μόνο τη πρόσφατου ισχυρισμού του Σνόντεν για κατασκοπίες και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, αλλά και του ε, παλιότερου ισχυρισμού πριν από πέντε χρόνια για υποκλοπές ε, στο Συμβούλιο Υπουργών στο κτίριο του Συμβουλίου Υπουργών ή παραβιάσεις του δικτύου στο κτίριο του ΝΑΤΟ. Είχαμε και τέτοιες καταγγελίες. Θεωρείτε ότι έχει ενισχυθεί η ασφάλεια και έχουν αποσοβηθεί τέτοιες επιθέσεις γιατί αυτό προσπαθούμε να ανακαλύψουμε στην έρευνά μας. Τι διασυνδέσεις ε, και τι σχέση υπάρχουν μεταξύ των παλιότερων καταγγελιών και των ε, τελευταίων, των πρόσφατων. Αν έχει ενισχυθεί η ασφάλεια, αν έχουμε καλύτερη δυνατότητα αντίδρασης σε τέτοιες ε, επιθέσεις. Δεν κάνουμε μια γενική και αφηρημένη έρευνα για το οργανόγραμμά σας ή το σχέδιο, το πρόγραμμα εργασιών σας. Μας ενδιαφέρει πώς ε, αντιδράσατε είτε γενικά είτε ειδικά ως προς αυτούς τους χειρισμούς και τις καταγγελίες. Και αν έχει ενισχυθεί η ασφάλεια των κοινωτικών θεσμικών οργάνων σε ό,τι φορά τα αισθήματα πληροφορικής μας. Ξέρω κύριε Πρίσο ότι δεν ε, μπορείτε να δώσετε πολλές πληροφορίες για την Βελγακόμ και μάλιστα στο παρελθόν σας είχαμε καλέσει, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσατε να έρθετε. Ξέρω ότι θα σας περιορίζει το απόρριτο, αλλά πείτε μας ό,τι ε, μπορείτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, ε, τη Eurodac, μας δώσατε κάποιες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις βελτιώσεις στο σύστημα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά πριν το καλοκαίρι ακούσαμε κάποιες καταγγελίες για παραβίαση του συστήματος SIS, του Schengen του, σύστημα πληροφο... συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Αυτά που μας είπατε ήταν ε, αντίδραση και διόρθωση αυτό που συνέβησαν το καλοκαίρι ή υπήρξαν ε, αποδείξεις για παραβίαση του συστήματος τακτυλικών αποτυπωμάτων, του συστήματος πληροφοριών του Σέγγεν ή όχι. Και αν ναι, τι κάνατε για να τις αποτρέψετε. Αυτά. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να μας πείτε τι συνέβη, πώς αντιδράσατε, πώς αντιμετωπίσατε τέτοιου είδους επιθέσεις και όχι μόνο αόριστα αλλά και πιο ειδικά. Ο κύριος Πρίντς πρώτα. Θα είμαι λακωνικός. Αν είχατε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για την Πελγακόμ θα έκανα μια απόπειρα να σας απαντήσω για να σας βοηθήσω. Αν μας κάνετε δύο ματιές είναι ναι, ε, τρεις ε, ναι, ε, δύο όχι. Θα σας κάνω νόημα με χαμόγελο. Ο κύριος Αμπαλιώνα. Το δεύτερο σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν δεν έχει υποστεί ε, παραβιάσεις. Ε, τον Απρίλιο είχαμε ε, μια καταγγελία για το πρώτο σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν όμως, που δεν υπόκειται όμως στην επιχειρησιακή διαχείριση του οργανισμού. Το νέο σύστημα ξεκίνησε τον Απρίλιο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μας ε, εκδηλώσαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κρούσμα, τα παραβίαση στο πρώτο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Βέβαια, το δεύτερο σύστημα ε, πληροφοριών Σέγγεν δεν έχει σχέση με το ΣΥΣ1. Αλλά το θέμα είναι τι μπορούμε να διδαχτούμε από το κρούσμα στο πρώτο ΣΥΣ. Τι κάναμε λοιπόν. αναγγέλαμε μια επανεξέταση end-to-end ε, για την ασφάλεια, μια ενδελεχή δηλαδή επανεξέταση του συστήματος και μάλιστα ο Επίτροπος ε, κάλεσε όλους τους επικεφαλείς ε, των αστυνομικών αρχών και συμφωνήσαμε να, να εκπονήσουμε ένα σχέδιο ασφάλειας μετά το κρούσμα στο ΣΥΣΕΝΑ για να δούμε αν το δεύτερο ΣΥΣ είναι ευάλωτο και έχει τα ίδια τροτά σημεία με το ΣΥΣ 1. Τα τροτά σημεία δηλαδή που εκμεταλλεύτηκαν οι hackers για να παραβιάσουν το πρώτο ΣΥΣ, το ΣΥΣ 1. Σήμερα προβαίνουμε σε μία ανάλυση των αποτελεσμάτων των απαντήσεων που μας έδωσαν τα κράτη-μέλη στο ερωτηματολόγιο που στείλαμε και θα κάνουμε τη συμπίληση αυτών των απαντήσεων και της ανάλυσης επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βό, ο πρώτος και ο δισηγητής. Ähm, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρίνς, θα ήθελα να επιμείνω, ίσως να το πω αλλιώς. Εγώ είχα διαβάσει πως υπήρχαν ίχνη ενδείξεις προς τη μεριά της Μεγάλης Βρετανίας ήταν σωστό ή όχι. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε ή όχι. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν θέλω να σας φέρω σε αμηχανία, αλλά ε, θα ήταν σημαντικό για εμάς να γνωρίσουμε, να γνωρίζουμε λίγο το, το υπόβαθρο της υπόθεσης. Ίσως βέβαια να ανακαιθεί τη ζήτημα επαγγελματισμού, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να το φτιάξει κάποιος μόνος του στον υπολογιστή του ή χρειάζεται κάποια εντατικότερη γνώση. Και κάτι άλλο θα ήθελα να γνωρίσω. Όλα αυτά τα οποία προέκυψαν μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιο συνδέθηκε πού και τι ε, πήρε και αν μπορούμε να το διαπιστώσουμε θα υπάρξει μεγαλύτερη επένδυση στην ασφάλεια θα απαιτηθεί περισσότερο ε, μεγαλύτερος προϋπολογισμός. Τι χρειάζεται για να είναι ασφαλής η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε βεβαίως οπωσδήποτε να βάλουμε μετά στις εκθέσεις μας, αλλά επίσης θα με ενδιέφερε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι βελτιώσεις και τι από αυτά μας αφορά και στην ε, καθημερινή μας λειτουργία. θέλετε να ακούσετε τις απαντήσεις ε, των τριών κυρίων. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Πρίντς. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ρωτήσατε για τη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίω είδαμε την ε, παρουσίαση που υπήρχε στο Σπίγκελ την Παρασκευή αυτό είναι το μόνο που έχω δει εγώ που σχετίζεται με τις, το αρχηγείο των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Τώρα, το τι προσπαθούν να κλέψουν επίσης μας δίνει μία ένδειξη για το ποιοι είναι οι δράστες αλλά αυτό πρέπει να γίνει βεβαίως ε, online και, και όχι εντός του δικτύου. Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται γιατί βεβαίως πρέπει να μπούμε εμείς σε άλλους υπολογιστές. Η άλλη ερώτησή σας για το επίπεδο. Η ίδια η ακόμη είπε πως ήταν πάρα πολύ πολύπλοκη και επαγγελματική επίθεση και ισχύει αυτό και νομίζω πως έπρεπε να φέρω και εγώ μία διαφάνεια ε, την απόφαση που πρέπει να λάβετε και πόσο θέλετε να επενδύσετε. Οι άλλοι, ας πούμε, εξοδεύουν δισεκατομμύρια. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσετε αν θέλετε να είστε σε θέση να υπερασπιστείτε αυτούς. και βεβαίως να διαλέξετε πού θέλετε να βρίσκεστε μετά ως διεθνής οργανισμός. Είναι δύσκολο να προστατευτείτε βεβαίως λόγω και της φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ο κύριος Ευχαριστώ. Το πρώτο που θα ήθελα να πω όπως είπα και στην εισαγωγή, είναι ότι συγκεντρώνουμε στατιστικές ε, για κρούσματα και ειδοποιήσεις ε, για παραβιάσεις και προσπαθούμε να αντιδράσουμε άμεσα. Δεν αναφέρθηκα σε συγκεκριμένα περιστατικά, γιατί δεν μπορώ να σας αποκαλύψω λεπτομέρειες για συγκεκριμένα περιστατικά. Μπορώ να απαντήσω μόνο γενικά τι έλεγχος έγινε για τους χειρισμούς που είδαμε στο ΔΥΠΟ ή αν ενημερωθήκαμε από εθνικές αρχές. Ναι, κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε την ελέγχουμε, τη διασταυρώνουμε, ελέγχουμε την ακρίβειά της και ελέγχουμε και τα δίκτυά μας. Και να φέρω και ένα παράδειγμα για την υπόθεση της Belgacom. Πριν από λίγες εβδομάδες ε, είχατε κρόση με τους εκπροσώπους της Belgacom που είπαν ότι έδειξαν, ε, έδωσαν κάποιους ε, δείκτες για το πώς ε, συνέβησαν αυτά τα περιστατικά στην πράξη και μάλιστα το έδωσαν μέσω της Fox IT και στη, τις έδωσαν και στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές και μάλιστα δόθηκαν αυτές οι πληροφορίες και στα εθνικέ ομάδες αντιμετώπισης εκτακτών αναγκών και στην Ευρωπαϊκή Ομάδα. Εμείς ελέγχουμε τις πληροφορίες όταν τις λαμβάνουμε και έχουμε επαφή με τους πολίτες, το Συμβούλιο, την ε, Επιτροπή, το Κοινοβούλιο. Έγινε λοιπόν ο έλεγχος ε, και η εξακρίβωση της, ε, των, στοιχείων, των στοιχείων αυτών και μετά από έλεγχο δεν βρήκαμε με τις τεχνικές πληροφορίες που είχαμε κάποια τροτά σημεία. Τώρα, κάθε φορά που είτε εμεί τα κοινωτικά θεσμικά όργανα ενημερωνόμαστε για μια πιθανή παραβίαση, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και να εντοπίσουμε αυτή την παραβίαση. Βέβαια, κάποιες παραβιάσεις τις εντοπίζουμε και από μόνοι μας στα δίκτυα, χωρίς πληροφορίες ή καταγγελίες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση γίνεται εκτενής έλεγχος και αν διαπιστώσουμε παραβίαση, τη διορθώνουμε το συντομότερο δυνατό. Τώρα, αν είναι δυνατόν να εντοπίσουμε αν έχει, υπάρχει wiretapping, παγίδευση ε, καλωδίων ή διαρροή πληροφοριών. Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς κάτι τέτοιο αν δεν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε ενδείξεις ότι κάτι πάει στραβά. Τότε μπορούμε να δούμε από πού διαρρέουν πληροφορίες. Πάντως γενικά είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί κάτι τέτοιο. Και να επαναλάβω αυτό που είπε και ο κύριος Πριντς. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν. Ακόμη και με τα πιο πρεγμένα μέσα να έχουμε 100% διαβεβαίωση ότι το σύστημά μας είναι αδιάβλητο απέναντι σε παραβιάσεις και επιθέσεις. Και η τελευταία ερώτηση, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να ενισχύσουμε την ασφάλεια προσπαθούμε κάθε φορά να αναβαθμίζουμε τις προδιαγραφές ασφάλειας και κάθε φορά που μαθαίνουμε κάτι από ένα κρούσμα ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε το επίπεδο προστασίας. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι δαπανηρό ε, και σε λογισμικό και σε αύξηση του προσωπικού. Είναι δαπανηρές αυτές οι ενίσχυσεις και αναβαθμίσεις της ασφάλειας. Επίσης, ε, ταυτόχρονα, Προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τη μόχλευση με τον καλύτερο συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και την καλύτερη διοργανική συνεργασία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολιτική υποστήριξη αυτή τη διοργανική συνεργασία, όπω είπε ο κ. Βιλέλα, για καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Κάτι τέτοιο είναι ευπρόσδεκτο. Και για να ολοκληρώσω, κάτι που προσπαθήσαμε σε κοινοτικό επίπεδο να εφαρμόσουμε ευθυγραμμίζεται και με την ευρωπαϊκή πολιτική για την υποχρεωτική ε, υποβολή εκθέσεων και την πολιτική της ασφάλειας στον κυβερνό χώρο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή να έχουμε αρμόδιες ομάδες που θα λαμβάνουν πληροφορίες για τα κρούσματα, τα περιστατικά παρεμβίασης και θα γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων φορέων των κρατών μελών. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε αρμόδια σώματα που μπορούν να αντιδρούν άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα. Ευχαριστώ. Κύριε Βιλέλα, έχετε να προσθέσετε κάτι. Oui, volontiers. Ναι, ευχαρίστω και σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω στην άμεση ερώτηση που έθεσαν οι τρεις ευρωβουλευτές. Τι κάνουμε καθημερινά και τι θα πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Καθημερινά προσπάθησα ακριβώς στην εισήγησή μου να σας υπογραμμίσω πώς εργαζόμαστε. Εμείς έχουμε μια παρακολούθηση καθημερινή και έλεγχο του τι συμβαίνει σε ολόκληρο το σύστημά μας. Και κάθε φορά που εντοπίζουμε κάποια προειδοποίηση, κάποιο συναγερμό, όπου μπορεί δηλαδή να φανταστούμε ε, ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάνουμε δύο είδους παρεμβάσεις. Μία άμεση για να δούμε αν ε, το πρόβλημα είναι πραγματικό και άρα μπορούμε να το λύσουμε άμεσα και η άλλη πιθανότητα είναι, δυνατότητα είναι να διευθυνθούμε στο ΣΕΡΤ ώστε να έχουμε μια πιο εις ανάλυση ενδεχομένως και με ε, κάποιες περισσότερες ενδείξεις. Ε, θα ακούσατε την έκθεση του κυρίου Τζαμπαλιώνε που μιλούσε για κάποιες προτάσεις για κριτήρια και μεθόδους και όταν μιλούσα για στάνταρ μεθόδους που ισχύουν ε, και εφαρμόζονται στην DG, DG e e ακριβώς περί αυτών πρόκειται. θα πρέπει να βελτιωθούν, αλλά πάντως αυτές τις γραμμές κινούνται. Για τα άλλα ερωτήματα ε, υπήρξε μια άμεση ερώτηση που αφορούσε την Πελγακόμα. Ναι, η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έχει κάνει μια εργασία εις βάθος ανάλυσης και στόχος ήταν να δει αν υπάρχουν ε, ε, υπάρχει αντίκτυπος για τα όσα συνέβησαν στη Βελγακόμ. Μπορώ να σα επιβεβαιώσω τώρα με κατόπιν ευρύτατη και δελεχούς ανάλυση ότι δεν ε, εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα ε, το οποίο να επηρέασε τις, ε, τα συστήματα του Ευρωκοινοβουλίου. Τρίτο ερώτημα, ε, αν πρέπει να επενδυθούν περισσότερα χρήματα. Ε, κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλα βήματα και να πάμε πολύ μακριά με τέτοιου είδους επενδύσεις. Θα πω επίσης ότι το επίπεδο των εμπειρογνωμόνων μας είναι εξαιρετικά υψηλό επί τη βάση ε, ε, διεθνών προδιαγραφών. Περισσότερες επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό το κεντρικότερο σημείο. Το κεντρικότερο σημείο, κατά τη γνώμη μου, είναι και η πρότασή μου είναι Τώρα, έπειτα είναι θέμα της Κομισιόν να δει αν θα το δεχτεί ή όχι. Να επιμείνουμε στα κεντρικά σημεία που ανέφερα στην εισήγησή μου την αρχική. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την διοργανική συνεργασία προχωρώντας περισσότερο στην ανταλλαγή πληροφοριών. Θα πρέπει να βρούμε συγκεκριμένες δράσεις, κοινέ δράσεις. Για παράδειγμα, δεν αρκεί, αλλά σίγουρα μπορεί να μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο των εξωτερικών δολίων πράξεων, το να φτιάξουμε δηλαδή μια κοινή δομή με κοινό ε, κύκλωμα, εντός του οποίου θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε μια ολόκληρη σειρά δομών. Και αυτό θα ήταν μια προληπτική ε, άμυνα και όχι διαδοχική. Σας ευχαριστώ και τώρα θα μιλήσω ως σκιώδηση της ομάδας μου, του Ισάλντε τον φιλελευθέρων. Θα ήθελα λίγο να εντείνω τη συζήτηση, γιατί ακούω ένα σωρό απαντήσει που λένε πολλά για διαδικασία και γραφειοκρατία, αλλά πολύ λίγα λέγονται για το τι συμβαίνει στην πράξη. σω αυτό να μην είναι εντυπωσιακό. Αν ακούσουμε ότι ο κύριο Πρίνς λέει πω η άλλη πλευρά, όποια και αν είναι, έχει δαπανίσει δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, ενώ εμείς έχουμε μια ομάδα, μια χούφτα στην ουσία ανθρώπους που πρέπει να οικοδομήσουν ε, άμυνα απέναντι στα δισεκατομμύρια, αυτή είναι χαμένη η μάχη από την αρχή. Και έχω και μια-δυο συγκεκριμένε ερωτήσει. Να αρχίσω με τον κύριο Πρίντ, που έχω μια ερώτηση σε σχέση με το SWIFT και έπειτα θα περάσω στην Πελγκακόμα. Μια απλή ερώτηση. Εσείς συμφωνείτε με την Ολλανδική κυβέρνηση πως η υποτιθέμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον σερβερ SWIFT στις κάτω χώρες μπορεί να ερευνηθεί σωστά χωρίς να γίνουν οι ε, ιατροδικαστικού τύπου ε, τεχνικές έρευνες. Πιστεύετε δηλαδή ότι η αρχή προστασία δεδομένων ε, μαζί, μαζί με την πελκική αντίστοιχη έχουν, είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για να κάνουν τέτοια έρευνα και να φέρουν στο φως την αλήθεια. Δεύτερη ερώτηση για την Belgacom. Η Belgacom μας είπε πως ε, πρόκειται για μαζική επίθεση ε, προηγμένου τύπου. Εσείς είπατε ότι δεν έχουν επηρεαστεί προσωπικά δεδομένα. Δεν έχουμε βρει ενδείξεις ότι έχουν υπάρξει υποκλοπές. Ο κόσμος ε, δαπάνησε εκατομμύρια εκατομμύρια, αλλά, αλλά δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί το σύστημα. Δεν μπορώ να τετραγωνίσω αυτό τον κύκλο. Κάτι λείπει εδώ. Γιατί θα, θα ε, έμπαινε κανείς τον κόπο να δαπανίσει εκατομμύρια εκατομμυρίων για να μην καταφέρει τίποτα. Μα δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Έπειτα ο κ. Δεζούρη είπε ότι δεν μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για την υπόθεση Μα Εγώ θέλω λεπτομέρειες, ιδιαίτερα γιατί μπορεί να έχει επηρεάσει το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα να καταλάβω, εσείς εντοπίσατε Εντάξει, αυτό που έγινε με την υπόθεση Μπέλγα, την ε, μάθατε πρώτα και μετά αρχίσατε να ερευνάτε. Ε, ήδη ανέφερα ότι είχαμε κάποιους ομιλητές της Microsoft, του Facebook, του Apple, ε, του Yahoo. Εσείς ακολουθείτε τα περιστατικά, τα κρούσματα της Belgacom. Έχετε δει πώς η Microsoft, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ανοίξει πίσω πόρτες, να είχαν δώσει τα συστήματά τους. Τι άλλο μας περιμένει. Πολύ συγκεκριμένα στον κύριο Πρίνς, γιατί είπατε ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε ίσως σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Υπάρχει κάτι που σας κάνει να πιστεύετε πως ε, το Ευρωπαϊκό μάλλον οι επικοινωνίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υποκλαπεί, έχουν παρακολουθηθεί ή εν πάση περιπτώσει τεθεί σε κίνδυνο. Αυτά. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά για την ώρα θα σταθώ σε αυτά. Και θα ζητήσω από τον κύριο Πρίνς να απαντήσει πρώτα και μετά θα ζητήσω από τον κύριο Ντεζούρε να απαντήσει. Σας ευχαριστώ. Πρώτη απάντηση. Ρωτήσατε αν μπορεί να γίνει μια έρευνα για να δείτε αν η NSA είναι εδώ πέρα. Μέσω κάποιων εγγράφων. Όχι. Πρέπει να δούμε τα συστήματα, τα τεχνικά. Δεύτερη ερώτηση ήταν το αν η ΣΕΜΠΕΠ, η υπηρεσία τεχνολογικής προστασίας της Ολλανδίας, ε, έχει επαρκείς πόρους. Ε, άκουσα χθε τον επικεφαλής να λέει πως θα προσλάβει νέο προσωπικό, οπότε αναγνωρίζουν πως χρειάζονται ε, και άλλους ειδικού. Τρίτη ερώτηση. Έχω γράψει εδώ πέρα ουδέν σχόλιο, αλλά δεν θυμάμαι ποια ήταν η ερώτηση. Ε, ναι, ταιριάζει σε πολλές ερωτήσεις το δεν σχόλιο. Εάν έχει... Ε, εάν ε, επικοινωνίες ή δεδομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υποκλαπεί κατά κάποιον τρόπο. Ναι, όχι, δεν θα απαντήσω. Να συγχωρείτε. Μάλιστα. Και η τελευταία ερώτηση. Έχει νόημα οποιοδήποτε φορέας να ξοδεύει δισεκατομμύρια όπως μας είπατε και μετά να μην υπάρχουν στοιχεία ε, παραβίασης. Ε, είναι λογικό αυτό? Εύκολα. Όχι. Δεν είναι λογικό. Μάλιστα, μα έλεγα, όπως μου φαίνονταν μόνο εμένα περίεργο. Κύριε Τιζέριο. Μάλιστα. Το ερώτημα σας ήταν ε, εάν ε, ανοιχνεύσαμε τα προβλήματα στην Belga.com. Η απάντηση είναι όχι. Αυτό σωστά εξήγησαν νομίζω πριν από λίγες εβδομάδες οι εκπρόσωποι της Belgacom. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν μόλις διαπιστώσαμε το συμβάν ήταν να ελέγξουμε εάν υπάρχει κάποιος αντίκτυπος στα θεσμικά όργανα. Και μπορώ να σκεφτώ δύο πράγματα. Το ένα ήταν μέσω του δικτύου της Belgacom ε, ήταν να έχει υπάρξει κάποια υποκλοπή των επικοινωνιών των βουλευτών ή του προσωπικού. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν έγινε κάτι τέτοιο ή όχι. Η Belgacom είπε πως ε, έχει υπάρξει, έχουν πληγεί τα δεδομένα των πελατών. Οπότε όπως ξέρουμε, ναι, δεν, έχει, δεν έχουν πληγεί, με συγχωρείτε. Οπότε, όπως ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν ε, έχει υπάρξει κάποια αποκλοπή δεδομένων ε, ευρωβουλευτών ε, ή προσωπικού. Κατόπιν, εάν το κακό λογισμικό επηρέασε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Με τα τεχνικά στοιχεία που έχουμε λάβει από τις έρευνες, δεν έχουμε βρει κάτι τέτοιο. Τώρα, πρέπει να πω πως Όλες αυτές ε, οι έρευνες ε, της περιπτώσεις ε, της Belgacom είναι επίσης στα χέρια της δικαιοσύνης, όπως ξέρετε, οπότε είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το να μιλάμε για αυτές τις υποθέσεις. Και είμαστε πολύ τυχεροί, θα έλεγα, για το ότι ο εισαγγελέα στην περίπτωση αυτή και η αστυνομία έχουν επιτρέψει σε εμά και κάποιους άλλους ε, να ελέγξουμε τα δίκτυα για το εάν είχαν επηρεαστεί ή όχι. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε πως είναι δύσκολο να δεχτείτε την απάντηση ουδέν σχόλιων. Η θετική πτυχή είναι πως μπορέσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα πρώτον και δεύτερον μπορούμε να σας πούμε με, κάποιο, με αρκετή βεβαιότητα πως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένδειξη για το ότι έχουν επηρεαστεί τα δίκτυα ή τα δεδομένα των θεσμικών οργάνων. Τώρα για αυτά τα οποία είπατε, Microsoft, Apple και ε, πιθανά παραθυράκια. Δεν γνωρίζουμε κάποια παραθυράκια τα οποία έχουν μπει εσκεμένα στο λογισμικό που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τώρα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Ειλικρινά δεν ξέρουμε. Ξέρουμε πως δεν έχουν μπει εσκεμμένα από τους πολιτές των προϊόντων. Τώρα ε, είναι ευάλωτα αυτά τα προϊόντα. Υπάρχει τρόπος να εισχωρήσει κάποιος σε αυτά τα προϊόντα οπωσδήποτε. ναι, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα η Microsoft ε, κάθε τρίτη βγάζει διάφορα patch ε, στους χρήστες για να κλείσουν ε, οι τρύπες. Και το Σαββατοκύριακο αυτό έγινε το ίδιο, μια πάρα πολύ σημαντική αδυναμία που ανακαλύφθηκε και είχε δημιουργήσει σούσουρο στον κλάδο μας καθώς μέσω του Internet Explorer ε, υπήρχε η δυνατότητα να πληγούν οι υπολογιστές των χρηστών. Ε, κάτι το οποίο ανακαλύφθηκε τη βδομάδα που μας πέρασε, έβγαλε το patch ε, αυτή την εβδομάδα η Microsoft. Βεβαίω, μάλλον το πρόβλημα, την αδυναμία αυτή την εκμεταλλεύονταν μήνες ή και χρόνια κάποιοι που το ήξεραν θα μπορούσαν τώρα αυτοί να είναι κράτη, ναι. Εγκληματίες, πιθανώς, ναι. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι πως δεν ξέρουμε, δεν έχουμε στοιχεία για το ότι αυτό ε, είχε γίνει από τους ε, είδους τους ε, κατασκευαστές του λογισμικού. Εμείς όμως πρέπει να φροντίσουμε να γίνουν αυτά στην ε, υποδομή που χρησιμοποιούμε για να είναι ασφαλή τα συστήματά σας. Σας ευχαριστώ. Έχω δύο ακόμη ομιλητέ σε αυτό το γύρο και ζητώ συγγνώμη από τους καλεσμένους ε, του δεύτερου πάνελ για τη μικρή καθυστέρηση. Ο Γιάνν Άλμπρεχτ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους ε, που δώσατε το παρόν στην ε, συνεδρίασή μας. Καταρχήν, στους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε ειδικευμένο προσωπικό για να κάνουν δοκιμές διείσδυσης στο σύστημα και πόσο συχνά γίνονται τέτοιες δοκιμές και πόσο συχνά αυτές οι δοκιμές έχουν θετικά αποτελέσματα. Εντοπίζω δηλαδή παραβιάσεις. Πόσα ακρούσματα έχουμε για επιτυχή παραβίαση συστήματος. Έχετε ειδοποιήσει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα ή άλλες αρχές ή φορείς ασφάλειας όπως η Βελγική Αστυνομία για πιθανές ε, κυβερνοεπιθέσεις προκειμένου να γίνουν σχετικές έρευνες από τις διεκτικές αρχές. Κύριε Πρίνς, μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι στις ε, Βρετανικές ε, αργίες και το μεσημέρι είχαμε σαφώς ε, χαμηλότερη δραστηριότητα των παραβατών, κάτι που ερμηνεύσατε. γιατί οι routers GRX είναι ιδιαίτερο στόχος των μυστικών υπηρεσιών ή πιο ευάλωτος. Και προς όλους τους καλεσμένους, τι έχετε να πείτε για τις επιθέσεις στην Belgacom πώς η υποδομή του Κοινοβουλίου ή των κοινοτικών θεσμικών οργάνων έχουν σχέση με την θηγατρική υπηρεσία της Belgacom. Θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους με τη σειρά που μίλησαν και στην αρχή. Κύριος Σπρίνς πρώτα. Και πάλι είναι δύσκολες οι ερωτήσεις. Δεν ξέρω, για τις αργίες και την ώρα του, τη μεσημεριανή διακοπή, δεν ξέρω και όσον αφορά το GRX ε, δεν ξέρω είναι ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρουσες ε, αυτές οι αδυναμίες για τις μυστικές υπηρεσίες. Κύριε Ντεζέρα, ούτε και εγώ έχω να προσθέσω τίποτα. Δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες για το τι μέτρα παίρνουν τα κοινοτικά θεσμικά όργανα για να προασπίσουν τα συστήματά τους. Μα εμείς είμαστε κοινοβούλοι, είμαστε ευρωβουλευτές, έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε αν ξεκίνησαν έρευνες από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα για πιθανές ε, επιθέσεις. Εσείς μας ρωτήσατε αν και πόσο συχνά κάνουμε δοκιμές διείσδυσης και πόσο συχνές, πόσο τι αποτελέσματα έχουμε, εμείς φροντίζουμε τα συστήματά μας να μην είναι ευάλωτα σε παραβιάσεις. Ε, εδώ δεν έχουμε μόνο συνομιλία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε και είναι δημόσια ακρόαση, μας ακούνε και πολίτες. Θα επαναλάβουμε την ερώτηση του κύριο Αν ζητήθηκε ε, δικαστική έρευνα. Για τι πράγμα λέει ο κύριος Ντεζούρα για πιθανέ κυβερνοεπιθέσει. Μα ρωτήστε με συγκεκριμένα. Ζητήθηκε έρευνα, να ζητηθεί δικαστική έρευνα με βάση πληροφορίες που βρήκαμε στον τύπο ή ε, κάτι που βρήκαμε στα δίκτυά μας. Έχουμε 40.000 ε, δελτία που παρουσίασε ένας, μια εφημερίδα μετά από στοιχεία που έδωσε ο Έντουάρτ Snowden υπήρχαν ειδοποιήσει ε, για κυβερνοεπιθέσει στα κοινωτικά θεσμικά όργανα και αν ναι, ενημερώσατε τι διοκτικέ αρχέ για να ξεκινήσει η δικαστική έρευνα. Αυτή είναι πολύ σημαντική πληροφορία για μα. Σας είπα, με βάση τις ε, πληροφορίε που είδαμε στον τύπο, ούτε η Κομισιόν ούτε κανένα άλλο θεσμικό όργανο έκανε καταγγελίες στις αστυνομικές αρχές. Ούτε νομίζω ότι είχε νόημα κάτι τέτοιο. όταν γίνονται καταγγελίες είτε στην αστυνομία είτε ζητείτε δικαστική έρευνα θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα κρούσματα, συγκεκριμένη παραβίαση, διάρρηξη, κλοπή. Δεν μπορούμε να ζητούμε έναρξη αστυνομική ή δικαστική έρευνα μόνο λόγω εικασιών ή πληροφοριών που κυκλοφόρησαν στι εφημερίδε ή στα μέσα μαζική ενημέρωση. Ο κύριο Βιλέλα, ευχαριστώ. Νομίζω ότι εγώ μπορώ να απαντήσω κάπω πιο ελεύθερα. Σε ό,τι αφορά Το εσωτερικό σύστημα τηλεφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πάροχος υπηρεσιών ε, είναι οι διατερία της τρεις έδρας του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνάψει συμβάσεις με την Belgacom, με την Orange και την Post του Λουξεμβούργου. Αυτοί είναι οι providers μας. Και φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται και από το δίκτυο αυτών των εταιριών και το εξωτερικό δίκτυο. Γιατί εμεί δεν μπορούμε να ελέγξουμε το εξωτερικό δίκτυο αυτών των εταιριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας, Interphone. Για αυτές τις εσωτερικές επικοινωνίες, όλα τα συστήματα που βρίσκονται είτε στο εσωτερικό ενός κτηρίου είτε μεταξύ συνδεδεμένων κτηρίων, όλο αυτό το σύστημα είναι κρυπτογραφημένο, ασφαλές και αδιάβλητο στις εξωτερικές επιθέσεις. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείτε το εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας ε, για να μιλήσετε μεταξύ σας ε, είτε στο, στο Στρασβούργο, είτε στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο. Αυτό το σύστημα το ελέγχει και το κρυπτογραφεί η Γενική Διεύθυνση ITEC. Και αυτό το σύστημα, επαναλαμβάνω, είναι αδιάβλητο. Σε ό,τι αφορά την προειδοποίηση, ναι, γίνονται καθημερινά έλεγχοι για πιθανές αδυναμίες και όταν εντοπίζουμε είτε κάτι συγκεκριμένο ή έστω και πιθανότητα παραβίασης, κοινοποιούμε την πληροφορία στην Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι και το όργανο που είναι αρμόδιο για περαιτέρω επεμβάσεις ε, και καταγγελίες είτε στην αστυνομία, μηνύσεις είτε ε, στα δικαστήρια προσφυγές. Εμείς ε, ε, εξασφαλίζουμε τις δράσεις στο πολιτικό επίπεδο. Και τρίτη δράση, εφαρμο... Ε, ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό ΣΕΡΤ, την Ευρωπαϊκή Ομάδα Κρούσης Εκτακτών Αναγκών, για να δούμε αν παρόμοια κρούσματα είχαμε και σε άλλα κοινωτικά θεσμικά όργανα, ώστε να οργανώσουμε άμεση αντίδραση παντού. Σας ευχαριστώ κύριε Ζαμπαλιώνε. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Αν έχουμε προσωπικό ειδικευμένο που να ασχολείται με τις δοκιμές διείσδησης. Ναι, φυσικά. Αυτό εμπίπτει στη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου. Θέλουμε πλήρη ασφάλεια του συστήματος. Έχουμε διάφορα μέτρα που εφαρμόζουμε ε, και εξακριβώνουμε την αποτελεσματικότητά τους με, την, με τον έλεγχο τροτότητας και δοκιμές δίδυσης. Μόνο έτσι είμαστε βέβαιοι αν είναι το σύστημα ασφαλές όπως ε, έχει σχεδιαστεί και αν μπορεί να παρέχει τις σωστές πληροφορίες. Τα συστήματά μας δεν είναι συνδεμένα με το διαδίκτυο και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Έχουμε κάποιες αρχές αυτοπροστασίας, ώστε ακόμη και τα δικτυά μας συνδέονται με εθνικά δίκτυα θεωρούμε ότι τα δίκτυα αυτά είναι αναξιόπιστα, ανάξια εμπιστοσύνη. Είχαμε ένα κρούσμα, επαναλαμβάνω, στο ΣΥΣ 1. Γι' αυτό και κάνουμε μια αναθεώρηση της ασφάλειας και του ΣΥΣ 2 και επίσης ε, μια δοκιμή διείσδυσης ε, στο ΣΥΣ 2 και μάλιστα σε κεντρικό επίπεδο για να διαπιστώσουμε αν το σύστημα το ασφαλές που ξεκίνησε τον Απρίλιο εξακολουθεί να είναι ασφαλές και προστατευμένο. Σε ό,τι αφορά τη, το νέο επιχειρησιακό μας δίκτυο, για την επικοινωνία μας και με τα άλλα θεσμικά όργανα και με το κοινό. Και για αυτό το δίκτυο έχουμε τις ίδιες αρχές πιστοποίησης της ασφάλειας με δοκιμές διείσδυσης και παραβίασης με τις οποίες δίνεται και τελική σφραγίδα και το πράσινο φως για την προστασία. Αν, δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα του τεστ διείσδησης, δεν πρόκειται να δοθεί το πιστοποιητικό ασφάλειας. Τελευταία ερώτηση για την κυρία, την Παρακαλώ να είστε σύντομοι, ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε σε 5, 6, 7 λεπτά και να προσπαθήσουμε έτσι να τηρήσουμε το πρόγραμμά μας. Όχι, έχουμε ήδη καθυστερήσει, αλλά πάση περιπτώσει να περιορίσουμε την καθυστέρηση. Κυρία Έρστε. Σας ευχαριστώ. Ε, τώρα συζητάμε τα δικά μας. Οπότε... Δεν ξέρω. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, ερωτήσεις και συμφωνώ με αυτό το οποίο υπόθηκε πως πρέπει να δούμε τα γενικά και δεν μπορούμε να δούμε τις ε, λεπτομέρειες. Ε, Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω και δεν μου επαρκεί αυτή η γενικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ξεκάθαρα το εξής. Γιατί βουλευτές, βοηθή, προσωπικό δεν έχουν αυτομάτως ένα κλειδί GPG. PGP μάλλον εννοεί η ομιλήτρια. Μπορείτε να μου Ισχύει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, το είπε ο κύριος ε, Τζεζερέ, πόσοι ασχολούνται στον τομέα της πληροφορικής. Εγώ θα ήθελα να μάθω πόσοι ασχολούνται ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ασφάλεια της πληροφορικής. Υπάρχει κανείς ή όχι. Αυτό προς τον κύριο Βιλέλα. Υπάρχουν εξωτερικοί ανεξάρτητοι έλεγχοι Γίνεται κάποιος έλεγχος διείσδυσης. Θα γίνει τώρα. Είναι πολύ αποφασιστικό αυτό νομίζω. Μετά. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάλι μπορείτε να αποκλείσετε πως ε, έχει υπάρξει ε, κάποια επίθεση στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για να διεισδύσει σε κάποιο άλλο θεσμικό όργανο. Μπορείτε να αποκλείσετε κάτι τέτοιο. Και ότι δεν είναι δυνατόν η κατασκοπία μέσω άλλου θεσμικού οργάνου. Επίσης τι κάνετε για να καλύψετε το κακόπιστο, το κακόβουλο λογισμικό. Μετά, εάν υπήρχε ας πούμε κάποια επίθεση ε, πώς θα μαθαίναμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει επίσης υποχρέωση ειδοποίησης και υπό ποιες συνθήκες θα ενημερώνονταν κάποια κοινοβουλευτική ομάδα ή ένας βουλευτής. Ποιες πληροφορίες υπάρχουν ακριβώς. Επίσης, η συνεδριαση κλεισμενων των θυρών που κάνουμε εδώ πέρα και βγάζουμε τον κόσμο έξω, πόσο ασφαλής είναι. Και εδώ πέρα θα ήθελα μία απάντηση. Είναι πολλές ερωτήσεις, το ξέρω. Θεωρώ πως μας οφείλετε απαντήσεις. Ναι, και είναι σημαντικέ ερωτήσει. Το θέμα τη ε, δοκιμή διείδηση ήδη ετέθη από τον Γιάννη Άλμπρεχτ. Δεν πήραμε πλήρη απάντηση και δεν νομίζω και ότι αν κάτσουμε εδώ περισσότερο θα πάρουμε περισσότερε λεπτομέρειε. Και επίση ε, κάποιε γενικέ ερωτήσει για την ασφάλεια που είναι σημαντικέ αλλά δεν έχουν σχέση με την έρευνα. Να εστιάσετε παρακαλώ στα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για την έρευνα μα. Ε, ερωτήσει βασικά τι κύριο Βιλέλα και στον κύριο Ντεζούρε. Κύριε Βιλέλα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ε, ναι, είναι όλες οι ε, ερωτήσεις εξαιρετικά ε, κερίες και σημαντικές. Όσον αφορά την ηλεκτρονική υπογραφή, εμείς, όπως γνωρίζετε, Πρόσφατα εισήγαμε την ε, ηλεκτρονική υπογραφή. Δεν ε, είναι ακόμα ένα μέσο που χρησιμοποιούμε. Ναι, το χρησιμοποιούμε μόνο για την ώρα σε πιλωτικό επίπεδο, δοκιμαστικά. δεν έχει ακόμα γενικευθεί η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής και ο λόγος είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι χρειάζεται να οριστεί το επίπεδο ασφαλείας που θέλουμε να επιβάλλουμε στην χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Όσον αφορά τα, τεστ διείσδυσης, Αυτά γίνονται διαρκώς. Και βεβαίως σε συντονισμό με το ΣΕΡΤΕ. Και εάν θεωρείτε πως ήταν σκόπιμο να γίνει ένα βήμα παραπέρα και να γίνει και έλεγχος εξωτερικού, εξωτερικός, πιστεύω πως ήταν καλή ιδέα. Ωστόσο, εμείς κάνουμε τακτικά δοκιμές για τα επίπεδα ασφάλειας και διείσδυσης του συστήματος. Αλλά δεν είναι εξωτερικός έλεγχος. Εγώ είμαι ανοιχτό και μάλιστα και ευνοϊκό στο να γίνει εξωτερικός έλεγχος για να δούμε ποιο να δούμε μάλλον πώς ε, θα γίνουν εξωτερικές δοκιμές, αλλά θα ήταν άχρηστο να μείνουμε στο επίπεδο του Κοινοβουλίου. Ένα τέτοιο πράγμα θα ήταν ε, χρήσιμο να γίνει με τα άλλα θεσμικά όργανα μαζί, τουλάχιστον τα δύο τα πιο σημαντικά που συνεργάζονται δηλαδή με το Κοινοβούλιο, που είναι η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Και αυτό μου επιτρέπει να απαντήσω επίσης στην τρίτη ερώτηση που θέσατε, δηλαδή εάν είμαστε βέβαιοι 100% ότι δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα από άλλα θεσμικά όργανα, να περάσουν μάλλον από άλλα θεσμικά όργανα για να μπουν στο δικό μας σύστημα για να επιτεθούν. Δεν είμαστε 100% βέβαιοι, όχι. Αλλά το σύστημα που φτιάξαμε με την δημιουργία του ΣΕΡΤ ακριβώς εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, να δίνει δηλαδή ε, συναγερμό και να προειδοποιεί. Και αυτό έχει γίνει συγκεκριμένα. Αν υπήρξε κάποιο περιστατικό σε ένα άλλο θεσμικό όργανο στην Κομισιόν, ε, το Κοινοβούλιο ενημερώνεται άμεσα, ειδοποιείται άμεσα ότι υπήρξε πρόβλημα και εμείς άμεσα ε, λαμβάνουμε τα μέτρα για να δούμε αν έχει γίνει του ίδιου είδους ε, επίθεση, αν θα μπορούσε μάλλον να γίνει του ίδιου είδους επίθεση και στο Κοινοβούλιο, ενάντια του Κοινοβουλίου. Και αυτό λειτουργήσε ως μηχανισμός προστασίας. Αλλά δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε 100%. Μπορείτε να ολοκληρώσετε. Ναι, αλλά μου, βάλ, μου θέσατε την ερώτηση. Το ξέρω, αλλά ε, δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Ντεζίρε, ναι, σύντομα για δύο από τα σημεία. Το ένα για την ε, κρυπτογράφηση του PGB. Δεν είναι πολύ εύκολο να να το εφαρμόσουμε. Το ζούμε καθημερινά ακόμα και στην επικοινωνία ανάμεσα σε, στους δεν είναι εύκολο να γίνει γρήγορα κρυπτογράφηση. Ε, θα ήταν ωραίο να είχαμε μια εύκολη λύση που θα προστάτευε τα email, τα τηλεφωνήματα ή τους φακέλους με κρυπτογραφημένο τρόπο. Και δεύτερο είναι πώς ανοιχνεύουμε τις ε, παραβιάσεις με διάφορα προγράμματα που έχουμε και software και πληροφορίες που λαμβάνουμε. Όμως τα περισσότερα τέτοια προγράμματα hardware και software και οι πληροφορίες και η ανταπόκριση στα κρούσματα είναι ε, εστιασμένη σε μια γεωγραφική περιοχή του κόσμου που δεν είναι η Ευρώπη. Αν δηλαδή ε, τη δική μου άποψη θα μπορούσα κάτι να προτείνω ως συμπέρασμα όλη αυτή τις συζήτηση σε αυτή την πολύ σημαντική επιτροπή είναι ότι οι τεχνικές λύσεις για την οργάνωση της κρυπτογράφησης για να έχουμε δηλαδή ασφάλεια για τα δίκτυα ε, και να έχουμε δηλαδή ανταπόκριση για να έχουμε ένα ασφαλές νέφος, όπως είπε και ο κύριος Ριβέλα πριν από λίγο, ε, όχι μόνο στο επίπεδο των θεσμών αλλά και στις χώρες μας, ε, με ευρωπαϊκές εταιρείες, ευρωπαϊκές λύσεις, αυτό θα ήταν σπουδαίο αποτέλεσμα. Θα μας βοηθούσε όλους αυτό στο μέλλον, νομίζω. Καλώς, σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το πρώτο τμήμα της συνεδρίασης με σχεδόν 20 λεπτή καθυστέρηση για την οποία και ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ τους καλεσμένους μας ε, από το πρώτο πάνελ για τις πληροφορίες τους. Σίγουρα θα αντιλήσουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, αν και έχω περισσότερες ανησυχίες τώρα από ότι στην αρχή της συνεδρίασης. Ε, δεν έχω καθυσυχαστεί καθόλου έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον προπολογισμό, γιατί ε, υφίσταται αλλεπάλληλε περικοπές αυτό ο προπολογισμό. Ενώ ε, οι εχθροί μα εντό εισαγωγικών ε, αυξάνουν τι επενδύσει του. Εμεί περικόπτουμε του προπολογισμού μα για την ασφάλεια. Ίσως θα πρέπει και εμεί να αυξήσουμε τις επενδύσει μας, αν θέλουμε κάπω πιο σοβαρή προστασία των συστημάτων μα. Θα ήθελα να καλέσω τώρα του καλεσμένου από το δεύτερο πάνελ Αλλάξε, παρακαλώ και τα ονόματα. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο τμήμα τη συνεδρία στο ρόλο τη κοινοβουλευτική εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο σε μια εποχή μαζική παρακολούθηση. Ε, τρίτο τμήμα. Ε, κοινοβουλευτική έρευνα 3, σαν το Ρόκι 3. Θυμίζει αυτές τις ταινίες που βγαίνουν σε πολλές ε, εκδοχές. Θα ήθελα, σε πολλές συνέχειες, θα ήθελα λοιπόν να περάσουμε στους τρεις καλεσμένους μας. Πρώτα θα ακούσουμε τις δικές τους παρεμβάσεις και μετά θα περάσουμε σε συζήτηση και ερωτήσεις. Θα καλωσορίσω πρώτα τον κύριο Αρμάντε Ντέκερ, που είναι αντιπρόεδρο τη Βελγική Γερουσία και μέλο τη Επιτροπή Παρακολούθηση τη Επιτροπή Εποπτεία των Μυστικών Υπηρεσιών. Και έχουμε δεξιά τον κύριο Πάχ... που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας των ε, Μυστικών Υπηρεσιών, γνωστή ως Επιτροπή R και ε, αριστερά του κύριο Κλοντ ε, Μωράς έχουμε τον κύριο Λάουριτσεν που είναι μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και εκπρόσωπος για θέματα νομικών υποθέσεων, κυβερνητικός εκπρόσωπος Εκπρόσωπο μάλλον τη της Βουλή, Βουλής, του Folketing. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για ένα δεκάλεπτο το πολύ με τη σειρά που τους παρουσίασα. Καλά μοιραστείτε εσείς μεταξύ σας το χρόνο και μετά θα έχουμε ε, ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο κύριος Ντεντέκερ πρώτα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας που στην ουσία αποτελεί συνέχεια των σχέσεων που υπάρχει ανάμεσα στη Βέλγιο και την Επιτροπή σας γιατί θυμάμαι πως είχα προσκληθεί ενώπιόν σας πριν από κάποια χρόνια με την ευκαιρία της έκθεσης που αφορούσε το Έσελον που ήταν η προηγούμενη φάση του προβλήματος που μας ε, απασχολεί σήμερα. Ε, Καταρχήν λοιπόν θα ήθελα εν συντομία να σας ε, εκθέσω πώς λειτουργεί το βελγικό σύστημα ελέγχου γιατί πιστεύω πως το σύνολο αυτού του προβλήματος συνδέεται και με τις ε, δυνατότητες ελέγχου με το τι, το τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες οι υπηρεσίες πληροφοριών των διαφόρων χωρών και θέλω να σας εξηγήσω πώς λειτουργούν όλα αυτά στο Βέλγιο. Σας θυμίζω το νομικό πλαίσιο που ξεκινά με ένα νόμο της 18ης Ιουλίου 1991. Ήδη δηλαδή έχουν περάσει 22 χρόνια οργανώνουν τον έλεγχο των ε, υπηρεσιών ε, πληροφορήσης, ναι, πληροφόρησης, μυστικών πληροφοριών και αστυνομικών αρχών. Πρόκειται λοιπόν για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τις μυστικές υπηρεσίες και τις αστυνομικές υπηρεσίες. Στο σημερινό πλαίσιο δεν θα αναφέρω βέβαια τον έλεγχο των αστυνομικών υπηρεσιών, αλλά μόνο τον έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών για να σας πω ποιος είναι ο ρόλος. Δηλαδή ασφάλεια, εθνική ασφάλεια πρόκειται για μια πολιτική υπηρεσία πληροφοριών και από την άλλη έχουμε και την ε, υπηρεσία των μυστικών πληροφοριών των ενόπλων δυνάμεων και έτσι έχει διοργανηθεί η μόνιμη επιτροπή ελέγχου των υπηρεσιών ε, πληροφοριών, η περίφημη επιτροπή ΕΡ, κομιτέ ΕΡ αποτελείται αυτή βασικά από την γερουσία. Με την μελλοντική εξέλιξη της γερουσίας θα είναι ε, το κοινοβούλιο που θα αναλάβει αυτή τη λειτουργία. Στη Γερουσία υπάρχει λοιπόν μια ειδική επιτροπή η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της Επιτροπής ΕΡ, της Κομιτέ ΕΡ και αυτή η Επιτροπή των Γερουσιαστών αποτελείται από πέντε γερουσιαστές και προεδρεύει αυτής ε, δικαιωματικά ο πρόεδρος της Γερουσίας. Αυτή η Επιτροπή εποπτεύει και συνοδεύει τη λειτουργία της Επιτροπής ΕΡ και η ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Παρακολούθησης ε, έχει τη δυνατότητα στο όνομα της Γερουσίας να αναθέτει στην Επιτροπή ΕΡ έρευνες, ε, να γνωρίζει όλες τις έκθεσεις, ε, ελέγχου που ασκεί η Επιτροπή ΕΡ, να τις κοινώνονται οι διάφορες έρευνες ώστε να επιτρέψει στο Γερουσία να προετοιμάζει πορίσματα και ενδεχομένω και συστάσεις. Η ίδια η Επιτροπή ΕΡ, κόμιτε ΕΡ, αποτελείται από τρία μέλη, τον Γενικό Εισαγγελέα κ. Ραπάη στα δεξιά μου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΡ, που ορίζονται από την Γερουσία τα τρία αυτά μέλη και αυτή η Επιτροπή ΕΡ επαληθεύει μέσω ελεγκτικών ερευνών αν οι ενέργειες μιας υπηρεσίας πληροφοριών έχουν θίξει με παράλογο ή άδικο τρόπο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων ή εάν διαπιστώνουν έλλειψη αποτελεσματικότητα συντονισμού. Από τη μια πλευρά έχουμε λοιπόν το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και από την άλλη την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αυτών. Μπορούν ε, να εκδώσουν μη δεσμευτική γνωμοδότηση για τις πολιτικές που πιστεύουν ότι είναι απαραίτητες ώστε να καλυφθούν ε, οι ελλείψεις, να προτείνουν συστάσει και ακόμα και να μετατρέψουν αυτές τις συστάσει σε προτα... νομοθετικές προτάσεις. Ε, αν αυτό χρειάζεται. Ω όργανο του Κοινοβουλίου, η Κομιτέ η Επιτροπή ΕΡ δεν έχει καμία ιεραρχική σχέση με τις υπηρεσίε πληροφοριών τις οποίες ελέγχει. Ε, δίνονται οι ε, διαβουλεύσεις στους αρμόδιους ε, ε, υπουργούς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Αμήνης και φυσικά ο Πρωθυπουργός αν αυτό είναι απαραίτητο και άλλες αρμόδιες αρχές ενδεχομένως ανάλογα με τους φακέλους όπως ας πούμε το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων σε ορισμένε περιπτώσεις που καταλήγουν σε, στα κατάλληλα συμπεράσματα ή λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Το Κοινοβούλιο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πορίσματα των ερευνητικών ελεκτικών των ερευνών για να προβεί σε νομοθετικές πρωτοβουλίες και για να ασκήσει το θεσμικό του έργο ελέγχου ε, επί της εκτελεστικής εξουσίας. Στο πλαίσιο της υπόθεσης Πρίσμα, η Επιτροπή Παρακολούθησης της Επιτροπής ΕΡ κάλεσε την Επιτροπή ΕΡ να ε, ξεκινήσει τρεις έρευνες ε, για τις οποίες θα σας ενημερώσει ο κ. Ραπάγη. Είναι προφανές ότι Κατά την άποψη της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής, η μαζική ε, παρακολούθηση επικοινωνιών από χώρες που θεωρούνται φίλες ή σύμμαχες έγινε υπό την ε, δικαιολογία της ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας, όμως τα μέτρα που λήφθησαν ήταν κατά τη γνώμη μας μέτρα τα οποία θίγουν τις βασικές αξίες, τις θεμελιώδεις αξίες που υποτίθεται ότι θέλουν να προστατεύσουν. Όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, φυσικά κανένας ε, καμιά, ε, δεν, ε, καμιά ενέργεια δεν δικαιολογείται από πλευρά των κρατών, δικαιολογείται η εποπτεία, αλλά όχι σίγουρα μια συλλογική και αδιάκριτη συλλογή στοιχείων. Όσον αφορά λοιπόν αυτήν την απίθανη μαζική παρακολούθηση των συστημάτων μας από τις αμερικανικές λέμε σήμερα υπηρεσίες, λέω πιθανή γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν θέλω να είμαι απόλυτα θετικός, όπως μάλιστα άκουσα και την, ε, ε, το, την ε, πρόνοια πολλών από τους όσους μίλησαν προηγουμένως, γιατί οι έρευνες, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί. Αυτές οι μαζικές παρακολουθήσεις έγιναν ίσως με τη βοήθεια ενός κρατούς μέλους της Ένωσης και αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο έχω την εντύπωση. Και άρα λοιπόν θεωρώ πως μια κοινή απάντηση σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν απαραίτητη. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να γίνει μεμονωμένα από κάθε κρατός μέλος. Επίσης θεωρώ ότι μια ανάλυση αυτής της κατάστασης ανάμεσα σε σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ, να θυμηθούμε ότι το ΝΑΤΟ είναι το κεντρικό μέσο ε, ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης, οφείλει και κατά την απόψή μου και το ΝΑΤΟ να ασχοληθεί με το θέμα και να ρυθμίσει το θέμα των σχέσεων ανάμεσα σε σύμμαχες φόρες. Διότι είναι πραγματικά αρκετά εντυπωσιακό ότι ανάμεσα σε συμμάχους ε, παρακολουθούμαστε. Αυτό που θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο επίσης και ίσως και να έχει ήδη ξεκινήσει θα ήταν αν κάποια κράτη-μέλη τη Ένωση διαπραγματεύονταν μια μεμονωμένη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Και γι' αυτό και μιλώ και για συζήτηση μέσα στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει φέρει σε δύσκολη θέση όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Προέρχεται ακριβώς από την ίδια διαδικασία που γνώρισα όταν ασχοληθήκαμε πριν από 10 χρόνια με το Έσελον, ότι δηλαδή πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης ασκούν δραστηριότητε τη ίδια φύση. Πρόσφατα άκουσα στην γαλλική τηλεόραση μια συζήτηση στην οποία συμμετείχε ο κύριος Αταλή ο κύριος Αταλή μιλούσε βεβαίως ε, προσωπικά, ονοματή του, αλλά έλεγε ότι με την εμπειρία του, γιατί ήταν για χρόνια γενικός γραμματέας του Ελίζε, Μπορώ να σας πω, έλεγε εκείνος, στους Γάλλους συναδέλφους που βρίσκονταν στην τράπεζα της συζήτηση ότι και η Γαλλία κάνει τα ίδια και ότι την είχε την δυνατότητα να κάνει περισσότερα, θα κάνει και περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. του θέματος ε, υποκλοπής ή παρακολούθησης. Μιλώ για τη Γαλλία, αλλά όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες κάνουν τα ίδια, σε διαφορετικά επίπεδα, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη κλιμάκια, εσελό. Ε, απάντως, ε, είναι αυτή η πραγματικότητα και θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθούν οι βασικές αρχές από κοινοβουλευτικές επιτροπές όπως σε τούτη εδώ και από κοινοβουλευτικές επιτροπές στα κράτη-μέλη. Θα σας θυμίσω ότι η πλειοψηφία των κρατών της Ένωσης δεν έχει ακόμα έλεγχο κοινοβουλευτικό επί των υπηρεσιών πληροφοριών τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και πιστεύω ότι ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις χώρες του ΝΑΤΟ κάποιοι κανόνες δεοντολογίας θα έπρεπε να υπάρχουν θα πρέπει επίσης να είναι ο κανόνας αυτός, χωρίς να είμαστε αγαθοί, αλλά προσπαθώντας να αποφύγουμε τις αποκλειστικές διμερείς συμφωνίες. Ήδη θα ήταν αυτό εις βάρος της πολιτικής αξιοπιστίας της Ευρώπης. Η διαπίστωση των υποκλοπών βεβαίως θα πρέπει να μας οδηγήσει να αναπτύξουμε ή να αποκτήσουμε μια ανεξαρτησία πληροφορική στην Ευρώπη. Το είπαμε πριν από λίγο ότι τα περισσότερα ε, πληροφορικά συστήματα που χρησιμοποιούμε δεν είναι ευρωπαϊκά. Με όλα όσα αυτά σημαίνουν, σημαίνει μάλλον όσον αφορά τους κινδύνους. Το ξέραμε όταν τα αγοράσαμε, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε αναπτύξει περισσότερα ε, συστήματα ευρωπαϊκά. Με πάνω από 500 εκατομμύρια κόσμο δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει. Αυτά είχα εγώ να σας πω και δίνω το λόγο στον κύριο Ραπάη. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ φυσικά να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας όπως και ο κύριος Ντέκερ και θέλουμε και ένα εθνικό όργανο ελέγχου να συμμετέχει στι εργασίε αυτέ και να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δύο υπηρεσίε πληροφοριών. Μία πολιτική που εξασφαλίζει την κρατική ασφάλεια. Πρόκειται για μια υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Και είναι μια υπηρεσία που ενεργοποιείται μόνο στο, στην Βελγική επικράτεια. Η δεύτερη υπηρεσία πληροφοριών είναι στρατιωτική και υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να δρά και εντό του Βελγίου αλλά και στην Ελλοδοπή. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο σε όλε τι χώρε. Μία, μία υπηρεσία πληροφοριών δεν έχει ούτε αστυνομικέ ούτε δικαστικέ δραστηριότητε. Ο έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών ασκείται κυρίω από την νομοθετική εξουσία και από την Ειδική Επιτροπή ε, Παρακολούθησης της Γερουσίας και την Μόνιμη Επιτροπή Επιτροπή Εποπτεία των Μυστικών Υπηρεσιών, την Επιτροπή ΆΡΟ, όπω περιέγραψε ο κ. Δεντεκέ. Η Επιτροπή μα απαρτίζεται από τρία μέλη, ορίζεται από τη Γερουσία και είναι σημαντικό αυτό ο συλλογικό χαρακτήρα τη Επιτροπή, γιατί εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τη Επιτροπή μα απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στου υπουργού, αλλά και απέναντι στι υπόλοιπε υπηρεσίε. Η Επιτροπή ε, έχει πολλά καθήκοντα, αλλά νομίζω ότι καλύτερα να περιστώ σε τρία που ενδιαφέρουν άμεσα την Επιτροπή σας. Καταρχήν, πραγματοποιούμε έρευνες ελέγχου, όπως λέμε στην δική μας ορολογία, είτε με δική μας πρωτοβουλία, είτε κατόπιν ετήσεως ε, του αρμόδιου υπουργού, είτε κατόπιν ετήσεως ε, του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Παρακολούθησης ή μετά από καταγγελία ενός πολίτη. Από τη δημιουργία της Επιτροπής μας πριν από 20 χρόνια, πάνω από 200 τέτοιες έρευνες ελέγχου έχουν διεκπαιρεωθεί. Μερικές μάλιστα από αυτές έγιναν για την υπόθεση SWIFT, για τις πτήσεις της CIA, το SLO, αλλά έγιναν και, έγινε και μια έρευνα για τις υποκλοπές στο κτίριο Just Lips του Συμβουλίου. Ο έλεγχος λοιπόν της Επιτροπής μας αφορά κυρίως την νομιμότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα και το συντονισμό του ελέγχου των υπηρεσιών πληροφοριών. Έτσι διαφοροποιούμαστε από αντίστοιχε υπηρεσίες των κατοχωρών για παράδειγμα γιατί εμείς πέραν της νομιμότητα ελέγχουμε και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Στόχος του ελέγχου είναι η πραγματοποίηση ενός ε, συνεχούς ε, δημοκρατικού ελέγχου που διαφυλάσσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, συμβάλλει όμως ταυτόχρονα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Δεύτερο σημαντικό καθήκον της Επιτροπής είναι η αρμοδιότητα που έχει από το 2003 και η δυνατότητα να ελέγχει τις παρακολουθήσεις ε, που γίνονται από τις στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες, Μάλιστα, οι στρατιωτικές υπηρεσίες, οι μυστικές, μπορούν να παρακολουθούν επικοινωνίες και στην Αλοδαπή, περιορισμένα όμως και να προστατεύουν τα βελγικά στρατεύματα που είναι αναπτυγμένα στο εξωτερικό και, καθώς, και επίσης τους βέλγους υπηκόους που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ε, εδώ και δύο χρόνια η υπηρεσία μας έχει και νομική αρμοδιότητα, οι υπηρεσίες έχουν την νομική αρμοδιότητα να κάνουν έρευνες σε ενδιαφέρουσες συχνότητες και μάλιστα η Επιτροπή μας προτείνει μετά από τη δίχρονη εφαρμογή αυτής της νέας αρμοδιότητας να διενεργήσει έλεγχο για το κατά πόσο γίνεται σωστή εφαρμογή της. Μια άλλη αποστολή της Επιτροπής είναι στα πλαίσια του νόμου για τις ειδικές μεθόδους συγκέντρωσης πληροφοριών. Οι βελικές υπηρεσίες από το 2010 έχουν ε, λάβει ε, ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων αρμοδιοτήτων, για παράδειγμα παρακολούθηση επικοινωνιών, συγκέντρωσης ε, τραπεζικών δεδομένων Οπότε η Επιτροπή μας ε, ε, λειτουργεί ως ε, ιδιάζων δικαστήριο. Έχει δηλαδή και δικαιοδοτικό ρόλο και μάλιστα σε οριστικό και τελεσίδικο βαθμό. Δεν υπόκεινται σε έδικα μέσα οι αποφάσεις μας. Εξετάζουμε περιπτωσιολογικά το σεβασμό από τις υπηρεσίες των αρχών της νομιμότητας, επικουρικότητας και αναλογικότητας. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι αρμοδιότητες που έχουν χορηγηθεί στις βελικές μυστικές υπηρεσίες με τον νόμο του 2010 αφορούν ε, επιχειρήσεις στη Βελγική επικράτεια και οι στόχοι θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένοι. Το ίδιο και οι απειλές θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, ειδικέ. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν επιτρέπονται στρατηγικές ή μαζικές παρακολουθήσεις όπως σε άλλες χώρες. Η Επιτροπή μας ανέλαβε και την διενέργεια τριών ερευνών από την Γερουσία και μάλιστα έχει προσθεθεί και μια τέταρτη έρευνα. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω το πλαίσιο αυτών των ερευνών, των τριών πρώτων και να πω και λίγα λόγια για την τέταρτη έρευνα. Η πρώτη έρευνα έχει τον τίτλο θα σας τον αναφέρω, ε, έρευνα ελέγχου για τη θέση των, υπηρεσι... των υπηρεσιών ε, πληροφοριών σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους ε, μαζικής συγκέντρωσης και επεξεργασίας μεταδεδομένων από κάποιες χώρες και τον τρόπο με τον οποίο χώρες αυτές ασκούν πολιτική κατασκοπία κατά δίθεν φύλων κρατών. Η Επιτροπή μας θα εξακριβώσει αν τι γνώριζαν ή τι δεν γνώριζαν οι βελγικές μυστικές υπηρεσίες ή τι όφυλαν να γνωρίζουν αν έδρασαν ενεργά στις άλλες χώρες ή αν δεν το έκαναν και επίσης αν ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές και μάλιστα εγκαίρως για τις πληροφορίες που έλαβαν. Είναι αυτονόητο ότι συνεχίζεται αυτή η έρευνα. Οι τελικές ακροάσεις ε, θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω πιο λεπτομεριακές πληροφορίες για το πέρας ε, και τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας. Γιατί ο νόμος μας υποχρεώνει πρώτα να υποβάλουμε τα πορίσματα της έρευνας αυτής στην Επιτροπή μας. Η δεύτερη έρευνα είναι νομικού χαρακτήρα, αφορά την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και των δεδομένων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή μας εδώ και πολλά χρόνια συστηματικά επιμένει στην ανάγκη να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των διαφόρων χωρών. Ε, δημοκρατικών χωρών θα ήθελα να προσθέσω εδώ. Τρίτη έρευνα που έχουμε αναλάβει στην Επιτροπή μας αφορά, με την, αφορά την προστασία του οικονομικού και επιστημονικού δυναμικού μας που μπορεί να υπονομευθεί από διάφορες ενέργειες παρακολούθησης. Ε, αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να σας το αναλύσω περαιτέρω. Η τέταρτη έρευνα ε, ξεκίνησε μετά από μια καταγγελία των Ολλανδόφωνων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Βρυξελών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι έρευνε ελέγχου, για τι έρευνε αυτέ, η Επιτροπή μα έχει σημαντικέ και εκτεταμένε αρμοδιότητε. Για παράδειγμα, συγκεντρώνει όλα τα κείμενα που χρειάζεται για να διεκπαιρεώσει την αποστολή τη. Έχει ακροάσει και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που κρίνουμε χρήσιμα για τι έρευνε. Δεν μπορούν μάλιστα να επεκαλεστούν επαγγελματικό απόρριτο για να αποκρύψουν πληροφορίε. Και επίση μπορούμε να κάνουμε κατάσχεση των χρήσιμων εγγράφων ή αντικειμένων για την έρευνα. Έχουμε και τα δικά μας αρχεία και επίσης ε, μπορούμε να ορίσουμε και ειδικού ή εμπειρογνώμονες για συγκεκριμένη έρευνα, όπως έγινε. Όπως είπα, ε, γίνεται μια πρώτη, ε, ένας πρώτος γύρος ερωτήσεων στείλαμε και ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο, συγκεντρώνουμε τα στοιχεία και τα τελικά πορίσματα θα οριστικοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε σε φάση συγκέντρωση πληροφοριών αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε σε θέση να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ε, με μια ιδιαιτερότητα. Όπως και εσείς και εμείς καθημερινά λαμβάνουμε νέες πληροφορίες και ε, διαβάζουμε νέες αποκαλύψεις. Αυτό που μέχρι τώρα ήταν μια εικασία μπορεί αύριο να γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο και κανείς δεν ξέρει. Τώρα, θα ήθελα να κάνω μερικές προτάσεις ε, για το πού θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει σημαντικό και πρωτοπόρο ρόλο. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των ελεκτικών οργάνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Οκτώβριο του 2010 έγινε στι Βρυξέλλε η έκτη διάσκεψη των οργάνων κοινοβουλευτικού ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα είχαμε συμμετοχή στη διάσκεψη αυτή της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Η διάσκεψη αυτή ολοκληρώθηκε με τη διακήρυξη των Βρυξελών και ε, το συμπέρασμα ήταν να αναγνωρίζουμε την ανάγκη και τη χρησιμότητα ανταλλαγής, ε, πιο έντονης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των οργάνων κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Βελγική Επιτροπή ανέλαβε και μια πρωτοβουλία δημιουργώντας ε, ένα ιστότοπο στο ΕΝΙΡ αλλά τα αποτελέσματα δυστυχώς, δυστυχώς υστερούν των προσδοκιών μας. Με εξαίρεση κάποιες συγκεκριμένες συνεργασίες μεταξύ κατοχωρών Γερμανίας και Νορβηγίας δεν έχουμε πιο εκτεταμένη συνεργασία όπως θα επιθυμούσαμε. Ωστόσο θα πρέπει να προβλέψουμε συγκεκριμένο προπολογισμό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ελεκτικών οργάνων. Άλλωστε αυτή ήταν η σύσταση και των καθηγητών Λί και Κάμερον την περασμένη εβδομάδα. Επίσης, αν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει την πρωτοβουλία μας για τον ιστότοπο ΕΝΗΡ είναι ευπρόσδεκτο. Δεύτερον, γνωρίζετε τον κανόνα της τρίτης υπηρεσίας. Έχει αναφερθεί συχνά αυτός ο κανόνας, είναι πολύ σημαντικός, αλλά θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εις βάρος ε, ενός ελεκτικού οργάνου. Οι εμπειρογνώμονες Λί και Κάμερον είπαν την περασμένη εβδομάδα ότι οι επόπτες δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τρίτη. Το βελγικό Ελεκτρικό όργανο ε, με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύει τον, τον κανόνα αυτό, φυσικά με την απαραίτητη σύνεση, ώστε να μην διακυβευτεί η ευρύθμη λειτουργία των βελγικών μυστικών υπηρεσιών. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι αυτό το θέμα συζητήθηκε και στην 7η διάσκεψη των ε, κοινοβουλευτικών οργάνων ελέγχου στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 2011. Και έκτοτε περιμένουμε πρωτοβουλίες που καλό θα ήταν να αναλυφθούν. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω τώρα να ακούσουμε τον κύριο Λάλτσεν από την Βουλή της ε, Δανίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ε, πρόσκληση λέει ο κύριος ε, Λάρτσιν, για να σας εξηγήσω ακριβώς το πώς λειτουργεί το δικό μας ε, το σύστημα και το τι έχουμε κάνει για τις υποκλοπές της NSA στην Δανία. Θα ήθελα λίγο σύντομα να πω κάποια πράγματα για τα δικά μας ε, τα ελεγκτικά όργανα και μετά να πω ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει το Κοινοβουλίο και η κυβέρνηση της ε, Δανίας. Πολλοί θεωρούν πως η Δανία είναι προοδευτική χώρα, αλλά όσον αφορά τον ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν είμαστε και τόσο προοδευτικοί, είναι λίγοι κοινοβουλευτικοί έλεγχοι μέχρι πρόπερση δεν είχαμε κάποια βάση. Τώρα έχουμε μια βάση για τον έλεγχο των ε, υπηρεσιών πληροφοριών και υπάρχει ανεξάρτητο όργανο εποπτείας τους. Ε, το όργανο όμως αυτό έχει πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες και εντολή. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε επιτόπου στις υπηρεσίες αυτές και επίσης ε, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε ακροάσεις ή τέτοια πράγματα, αλλά δεχόμαστε τις καταγγελίες ε, των πολιτών και βλέπουμε τι έχει γίνει και αν υπάρχει σωστή διαχείριση των δεδομένων τους. Χοντρικά αυτά μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει εδώ και χρόνια Και επίσης η Επιτροπή ε, Ελέγχου στο Φολκέτινγκ, την Βουλή της Δανίας, οι οποίοι είναι οι μόνοι που είναι σε θέση να έχουν διάλογο με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Όπως είπα, η Επιτροπή υπήρχε πολλά χρόνια, αλλά πέρσι ξεκαθαρίσαμε μετά της νομικής βάσης. Οπότε, όπως είπα, η Επιτροπή δεν μπορεί να κινητοποιηθεί ευθορμήτως, λαμβάνει στατιστικά προϋπολογισμούς και κοιτάει αν είναι αναλογικά, αλλά δεν εποπτεύει πλήρως τις υπηρεσίες ε, ασφαλείας. Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα να διαβιβαστούν πράγματα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και τώρα όσον αφορά την ε, συζήτηση την επίκυρη. εμείς επικεντρωθήκαμε κυρίως στην προστασία των δεδομένων. Εάν δούμε δε την εμπιστοσύνη που υπάρχει, αυτή προς τις υπηρεσίες ε, πληροφοριών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και στις περισσότερες, ε, περισσότερες περιπτώσεις ε, δικαίως. Ε, ίσως να είναι και υπερβολική εμπιστοσύνη, δεν ξέρω. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται όπως είπα με την προστασία των δεδομένων, όχι μόνο λόγω των αποκαλύψεων ε, Snowden, και των υποκλοπών π.χ. στο τηλέφωνο της ε, κυρίας Μέρκελ, αλλά είχαμε και άλλη μια περίπτωση στη Δανία, ένας Σουηδός χάκερ και ένας νεαρός Δανός χάκερ είχαν πρόσβαση σε πάρα πολλά δεδομένα επί σειρά των χωρίς να το έχει αντιληφθεί κανείς. Η μηνών, με συγχωρείτε π.χ. στα συνθηματικά του email ολόκληρης της αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτές τις πληροφορίες. Τελικά αποκαλύφθηκαν, συνελήφθησαν, δεν υπήρχαν ξένες δυνάμεις, ούτε επαγγελματίες hacker. Ένας νέος ήταν Μπήκε σπίτι του η αστυνομία, ήταν ξυπόλυτος στο κομπιούτερ. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και μετά η υπόθεση των υποκλοπών της NSA και των παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα το αξιόλογο, δεν ξεκίνησε κάποια έρευνα. Και μάλιστα μας είπαν πως σύμφωνα με τα όσα ξέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν υπήρχε παρακολούθηση κανενός ε, Υπουργού της Δανίας. Πώς το διαπίστωσαν αυτοί δεν ξέρω. Μας είπαν ε, έτσι έχουν τα πράγματα. Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων είπε πως το διαπιστωσαν αυτοι δεν ξερω μας ειπαν ετσι εχουν τα πραγματα η αρχη προστασιας προσωπικων δεδομενων ειπε πως θέλει να περιμένει, αναμένει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν κάνει κάτι παραπέρα. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, να συνεργαστεί με άλλες υπηρεσίες για να δει τι γίνεται στην περίπτωση της NSA και τώρα θα δούμε εάν ε, υπάρχει νομική βάση για αυτά τα οποία ζητήθηκαν. Και η Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ε, το τι θα κάνει από εδώ και μπρος ε, είναι ανοιχτό. Γιατί όπως είπα ό,τι γίνεται είναι εμπιστευτικό και δεν μπορούν να μας πούν το τι κάνουν, το τι γνωρίζουν καμία πληροφορία δεν μπορεί να βγει προς τα έξω. Υπάρχει λοιπόν τώρα πολύ μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση της Δανίας για να προχωρήσει σε βάθος, να δει πώς θα συνεργαστεί με άλλες υπηρεσίες και πώς θα προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών που κινούνται στο διαδίκτυο. Επίσης ασκήθηκε κριτική στο ότι ο Πρωθυπουργό και Υπουργό Δικαιοσύνη προσπάθησαν να κάνουν κάτι το οποίο ε, δεν ήταν απολύτως ε, σωστό. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια και δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι ως προς αυτό. Τέλος πάντων τώρα αυτό είναι το σύστημα που έχουμε και στο σύστημα της Δανίας όπως είπα δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό έλεγχο επί των υπηρεσιών ε, ασφαλεία. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε θέλουμε ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο ή όχι. Παριστάνουμε πως υπάρχει έλεγχος, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα. Και σε σχέση με αυτές τις ε, αποκαλύψεις. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής το Κοινοβούλιο έχει επικεντρωθεί ίσως το ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, πρέπει κάποιες δραστηριότητες να σταματήσουν. Πέρσι είχαμε 810 δισεκατομμύρια ξεχωριστά στοιχεία ε, δεδομένων που συλλέχθηκαν στη Δανία από το ίντερνετ ε, και δεν υπάρχει καμία αναλογικότητα με το τι χρειάζεται η αστυνομία για να καταπολεμήσει ε, την τρομοκρατία ή οτιδήποτε άλλο θέλει να καταπολεμήσει το ίντερνετ. Η τρομοκρατία δεν υπάρχει πάρα πολύ. Υπάρχει βεβαίω πολύ οργανωμένο έγκλημα. Ε, οπότε τίθεται ένα ζήτημα αναλογικότητας αλλά τέλος πάντων όπως σας είπα η συζήτηση αυτή σχετίζεται άμεσα με τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα προχωρήσει στην Δανία πριν προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε Μπορούμε, όπως είπα, να κάνουμε κάποια πράγματα στα εθνικά κοινοβούλια, αλλά θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρξει κάποια αποτελεσματική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μια... Υπάρχουν νομίζω κάποιες λογικές πρωτοβουλίες ε, που αφορούν τον νέφος, το λεγόμενο του διαδικτύου, η πρωτοβουλία για το διαδίκτυο, πρέπει να υπάρχει μια λογική προστασία των προσωπικών δεδομένων και των όσων συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Αυτή ήταν η δική μου τοποθέτηση. Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Λάουριτσαν. Περνάμε τώρα στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Κάποιοι συνάδελφοι έφυγαν και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ε, είμαστε και στο τέλος της εβδομάδας και προσπαθούν βεβαίως να προλάβουν και το αεροπλάνο. Θα ζητήσω τώρα τον κύριο Κλοντ Μωράες να μας πει κάποια πράγματα. Πράγματι σας ευχαριστώ για την πολύ αναλυτική παρουσίασή σας. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε το τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος και να το αξιολογήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους ε, συναδέλφους από τη Βελγική Γερουσία να ξεκαθαρίσουν το εάν η Βελγική Επιτροπή Εποπτείας μπορεί να δει της ε, διεθνής ε, τις ε, διεθνείς συναλλαγές που υπάρχουν. Δηλαδή, όπως μας είπατε, υπάρχει δυνατότητα διερεύνησης ατομικών καταγγελιών. Αυτό το οποίο περιγράψατε είναι ένα πάρα πολύ λεπτομερές σύστημα και υπάρχει κάποια διαφάνεια, αλλά το ερώτημα είναι αν σε εμποδίζει ο κανόνας του τρίτου μέρους. Όταν ξέσπασε η υπόθεση PRISM, θεωρήσατε πως α, οι διατάξεις που υπήρχαν για την υποπτία μαζί με τα όσα ακούστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το SWIFT και δεδομένου του ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βρίσκονται στο Βέλγιο, θεωρείτε πως αυτά τα οποία έχετε ε, παρκούνι, ότι χρειάζεστε κάποια μεταρρύθμιση, γιατί τώρα ακούμε από διάφορα κράτη-μέλη ε, πως έχουν κάποια συστήματα εποπτείας, τα οποία χρειάζονται μάλλον μεταρρύθμιση, οπότε ως ε, βουλευτές μάλλον είχατε κάποια εμπειρία. Πείτε μας λοιπόν, θεωρείτε πως υπάρχει επαρκής ε, εποπτεία ή εμποδίζεται από τον κανόνα του τρίτου μέρους και για τον συνάδελφο από τη Δανία. Είχαμε επίσης στοιχεία από Σουηδούς βουλευτές αρμόδιους για την Επιτροπή Εποπτείας και προφανώς ε, υπήρχαν ε, κατηγορίες κατασκοπία ει βάρος άλλων σκανδιναβικών χωρών της Δανίας. Δεν ξέρω αν το είπατε. Είπατε πως βεβαίως ε, δεν υπήρχαν πολλές τέτοιε κατηγορίες τέτοιε στην ε, Δανία. Οπότε σαφώς ε, είπατε πως δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία. Αν ισχύει κάτι τέτοιο βεβαίως για μια τέτοια περίπτωση θα, ε, θα είχε κινήσει το ενδιαφέρον. Υπάρχει κάποια δημόσια συζήτηση για την βελτίωση της εποπτείας στην Δανία. Εάν ναι, ακολουθείτε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, ακολουθείτε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό κράτος, ένα σκανδιναβικό μοντέλο. Εμείς θέλουμε να εστιάσουμε σε μια καλύτερη υποπτία δεδομένων των πάρα πολλών κατηγοριών που ακούγονται τώρα πια. Θα ήθελα λοιπόν την, την άποψή σας. Καθώς νομίζω πηγαίνετε προς ένα νέο σύστημα υποπτίας. Σας ευχαριστώ Κλοντ. Ήθελα να ζητήσω τους ομιλητές μας να απαντήσουν με την ίδια σειρά όπως πήραν το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος και ο κύριος Ραπάη θα συνεχίσει για τα μέσα που έχουμε σε σχέση με αυτά τα σημαντικά διεθνή φαινόμενα, θα έλεγα πως διαπιστώνουμε πως όταν ξέσπασε η υπόθεση Έσυλων πριν από 10 χρόνια, μόνο δύο κοινοβούλια έκαναν έρευνα. Το Γερουσία, η Βελγική, η Επιτροπή μας και το Ευρωκοινοβούλιο. Ήμασταν οι δύο και μοναδικοί. Και είναι προφανές ότι όταν κάνει η Επιτροπή αυτή την έρευνα, την κάνει ε, στις ε, υπηρεσίε πληροφορίες βέβαια. Βέβαια κάποιες πληροφορίες στάνουν στις επιτροπές που βεβαίως πάντοτε πρέπει να διαλέξουν τι μπορούν να πούν και τι όχι. Διότι στα θέματα πληροφοριών ε, το απόρριτο της πηγής είναι βασικό στοιχείο. Πάντως πιστεύω ότι με αυτού του είδους την εργασία, όπως κάνουμε και για το πρίσμα, αυτό θα εξοπλίσει την βελγική κυβέρνηση στην διεθνή της δράση και στα διεθνή φόρα, ώστε να μπορεί να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν κανείς δεν είναι καλά ενημερωμένος δεν μπορεί να πει τίποτα σωστό και φοβάται μήπως γελιοποιηθεί. Και όσον αφορά τα άλλα νομικά και τεχνικά ζητήματα, ο κύριος Ραπάγη ίσω είναι ο καταλληλότερος για να απαντήσει. Ναι, εγώ θα σα εξηγήσω με δύο λόγια τις αρμοδιότητε της Επιτροπής. Το νομοθετικό οπλοστάσιο είναι επαρκές, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μα πως η αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να παρακολουθήσει τι βελγικές υπηρεσίε τις βελγικές και μόνο αυτές. Δεν έχουμε αρμοδιότητες για τις ξένες υπηρεσίες που είναι παρούσες στο Βέλγιο και ενεργές στο Βέλγιο. Πέρυσι, μετά από αίτημα του προηγούμενου Προέδρου της Γερουσίας μάλιστα, μια έρευνα που αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο οι βελγικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τις ξένες μυστικές υπηρεσίες που δρούσαν στο Βέλγιο όταν αυτές ήταν αρκετά εκτεταμένε στο Βέλγιο. Θα προσπαθούσαμε να δούμε δηλαδή πώς λειτουργούσαν οι βελγικές υπηρεσίες εποπτεύοντας τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι ξένες αυτές υπηρεσίες είναι φίλες εντός εισαγωγικών, τουλάχιστον αυτές που είναι, έχουν σημαντική παρουσία στην επικράτειά μας. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή ότι Πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε τις φίλες ξένες μυστικές υπηρεσίες που είναι στο Βέλγιο. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο διότι υπάρχουν και ξένες και μάλλον και εχθρές υπηρεσίες ε, στις Βρυξέλλες. Ε, πρέπει δηλαδή με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να προσπαθήσουμε να θεσπίσουμε προτεραιότητες. Εμείς ζητάμε και πολλά χρονχή. Ε, συμπεριληφθεί στην νομοθεσία μας. Θα ήταν ίσως μια απαραίτητη αλλαγή που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ζητήσαμε στην νομοθεσία περί μυστικών υπηρεσιών να αναφέρεται ρητά πως οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των μυστικών ξένων μυστικών υπηρεσιών στην ευελική επικράτεια, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι στο πλαίσιο αυτό. Οι δυνατότητες της επιτροπή είναι αρκετά περιορισμένες. Είμαστε τρία μέλη. Δεν είμαστε μόνο τρεις, γιατί έχουμε και μια ερευνητική υπηρεσία και μια νομική υπηρεσία και μια υπηρεσία τεκμηρίωσης καθώς και δικαιωτική στήριξη. Είμαστε περίπου 25 άνθρωποι δηλαδή για να ελέγχουμε τις βελγικές υπηρεσίες που έχουν πολλά να κάνουν, ιδιαίτερα εδώ στις Βρυξέλλες. Εκεί που υπάρχει ένα εξαιρετικά λεπτό θέμα είναι το τεχνικό θέμα. Όταν μιλάμε για πληροφορική, πρέπει να έχουμε ειδικού ε, ε, εχμής, εμπειρογνώμονες και οι επενδύσει είναι σημαντικές. Το Βέλγιο, όπως και πολλές άλλες χώρες, αντιμετωπίζει, όπως και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοσιονομικές δυσκολίες, πράγμα το οποίο δεν ε, είναι καλός ιονός για τη συνέχεια θα δοθεί τα επόμενα χρόνια και πιστεύω πως αυτό θα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Οι επενδύσεις δηλαδή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την προστασία των υποδομών, το, της πληροφορικής εδώ στο Βέλγιο. Υπήρξε μια απόφαση της κυβέρνησης που ελήφθη μάλιστα μετά από μια σύσταση του 2011 και η κυβέρνηση το συμπεριέλαβε στην ε, κυβερνητική της δήλωση του 2011 αλλά και μετά από τα πρόσφατα γεγονότα Σνόντεν κτλ. Ε, πήρε την απόφαση να επενδύσει σχετικά μεγάλα ποσά για την προστασία του δικού του κυκλώματος ε, πληροφορικής, ε, πράγμα που είναι μια αρχή. Είμαι όμως πάντα αρκετά επικριτικός γιατί πολλά χρόνια η, Ευρωπαϊκή, η Βελγική Επιτροπή Ελέγχου των Μυστικών Υπηρεσιών ζητούσε να πάρει τέτοια μέτρα η κυβέρνησή μας και χρειάστηκε να περιμένουμε αυτή την υπόθεση Snowden ώστε επιτέλους να απεμπλακούν τα πράγματα σε ε, δημοσιονομικό και πολιτικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόριτσεν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά το δανέζικο σύστημα, όπως σας είπα, τον περασμένο χρόνο κάναμε ένα μικρό νόμο. Και από την πλευρά λοιπόν των μυστικών υπηρεσιών, η Επιτροπή Δικαιοσύνης μας έκανε ένα ταξίδι στην Ορβηγία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και έπειτα γινόταν δουλειά για 10 χρόνια και οι συστάσεις τους κατέληξαν στο εξή. Στο, μάλλον σε αυτή την νομοθεσία που πέρασε πέρυσι. Και Τώρα γίνεται συζήτηση για να φτιάξουμε μια νέα νομοθεσία και όπως αν τώρα γινόταν νέα νομοθεσία θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα λόγω της υπόθεσης Σνόντεν. Αλλά πέρασε ήδη πέρσι και δεν υπάρχει πολιτική πίεση για να αλλάξει αυτή η νομοθεσία. Ακόμα και αν γίνονται κάποιες συζητήσεις και κοινοβουλευτική συζήτηση, δεν νομίζω πως θα αλλάξει τώρα κοντά η νομοθεσία ώστε να δώσει περισσότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο ή νομικό έλεγχο στις ε, μυστικές υπηρεσίες μας. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Για τη Σουηδία ε, υπήρξε κάποια συζήτηση στην ε, Σουηδία για την δανέζικη περίπτωση, η Σουηδία παρακολουθεί όλα όσα μπαίνουν στο σύστημά της, αλλά και όσα βγαίνουν. Δηλαδή, αν εγώ, ε, αν ας πούμε το facebook μου μάλλον το σερβερ του facebook μου ε, πήγαινε εκεί, θα μπορούσε η Σουηδία να ελέγξει ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει από το σύστημά της. Όπως καταλαβαίνετε όμως δεν υπάρχει πολιτική πίεση στην κυβέρνηση, υπάρχει κοινοβουλευτική συζήτηση, αλλά δεν είναι σε τόσο ψηλό επίπεδο. Και υπάρχει μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης στις μυστικές μας υπηρεσίες και αυτό είναι μια βάση, υπάρχει βάση μάλλον για να έχουμε εμπιστοσύνη. Αλλά Μπορώ να σας δώσω ένα σύντομο παράδειγμα. Νομίζω πως αν και η παράθεση που θα κάνω, αν αυτό προερχόταν από κάποιον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε μια άλλη ευρωπαϊκή ε, χώρα, ε, θα γινόταν συζήτηση στα ΜΜΕ. Πάντως, ένας Δανός ε, βουλευτής είπε, σε σχέση με τον ΕΣΕΙ, ότι καταλάβαινε απόλυτα καλά γιατί ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί για την Ευρώπη, γιατί εμεί δημιουργούμε πολλά προβλήματα και ότι αν ήταν Αμερικανό και αυτό θα κρυφάγκουγε για τους δεν ήταν εστιάκι, το είπε σοβαρά. Αλλά δεν δημιουργήθηκε καν μια φασαρία για αυτά τις δηλώσεις. Η Δανέζικη κοινή γνώμη και η συζήτηση περί έλλειψης ε, ιδιωτικού χώρου και ιδιωτικότητας στη Δανία δεν υφίσταται. Είναι κάπως, ε, ε με φοβίζει κάπως αυτό πρέπει να πω, αλλά πιστεύω πως το εγγύς μέλλον θα αλλάξει. Πάντως για την ώρα, όπως σας είπα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της προστασίας των δεδομένων στη Δανία. Ευχαριστώ. Τώρα μιλώ και ως Πρόεδρος, αλλά ως και οδησηγητρία των φιλελευθέρων. Ε, θα γίνω εδώ ο δικηγόρος του διαβόλου, γιατί συνεχίζεται η έρευνά μας. Και ανήκουμε στην ίδια πολιτική οικογένεια. και το κόμμα σας συμμετείχε και σε προηγούμενες κυβερνήσεις ε, και συμμετείχε στην έγκριση νομοσχεδίων. Η Δανία, όπως και κάτω χώρες, αναφέρονται ως τέσσερις βασικές χώρες σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι συμπατριώτης σας. Διαρωτώ με λοιπόν αν νιώσετε πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Δανία για να αποφύγετε πιο αυστηρούς μηχανισμούς εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών και αν όχι πίεση έστω φιλική παρένεση να γίνει κάτι τέτοιο. Προς τους Βέλγους καλεσμένους μας θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε κι εσείς ε, στο θέμα αυτό. Πόσα ήξεραν οι μυστικές υπηρεσίες, ε, τι, ήξερα, τι γνώριζε η κυβέρνηση και σε ποιο βαθμό οι μυστικές υπηρεσίες ε, αυτενέργησαν. Έχω όλο και περισσότερες απορίες και ερωτηματικά Μήπως οι μυστικές υπηρεσίες ελέγχουν τις κυβερνήσεις. Γιατί προβληματιστήκαμε και με τη Γερμανία. Τι γίνεται αν έχει παγιδευτεί το κινητό τη καγκελαρίου. Το γνώριζαν αυτό οι μυστικές υπηρεσίες. Αν το γνώριζαν σημαίνει ότι είναι τελείω ανίκανε. Ή μήπως γνώριζαν την παρακολούθηση και δεν την ενημέρωσαν ή μήπω την ενημέρωσαν και εκείνη δημοσίω έκανε πω δεν το γνώριζε. Υπάρχουν πολλέ πιθανότητε εδώ, πολλά σενάρια. Τι συμβαίνει στο Βέλγιο, γιατί αν όλε οι μυστικέ υπηρεσίε, ε, τα έκαναν πλακάκια με τι αμερικανικέ και ποιο ξέρει με ποιον άλλον, ε, σημαίνει ότι οι μυστικέ υπηρεσίε του Βελγίου γνώριζαν την κατάσταση και σα την απέκρυψαν εμένα. Ή μήπω είναι το αντίθετο. Μήπως ε, οι διαδοχικές κυβερνήσεις έδιναν σχετικές εντολές στις μυστικές υπηρεσίες για συνεργασία. Τι γίνεται με τις βελικές μυστικές υπηρεσίες, είναι εκτός του παιχνιδιού ή μήπω είναι μέσα στο παιχνίδι, μέσα σε αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία. Οπότε αυτοί οι μηχανισμοί εποπτείας που έχετε, που φαίνονται αρκετά αποτελεσματικοί για αυστηροί, πώς δεν κατάφεραν να να εντοπίσουν τέτοιες παραβιάσεις. Σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα. Μπορεί να έχουμε εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας και μάλιστα ισχυρούς. Σε άλλες χώρες έχουμε πιο ασθενείς ε, ε, μηχανισμούς εποπτείας, αλλά ε, όπως σε όλες τις αλυσίδες, ε, η αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος της ε, κρίκος. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχουν πιο ασθενείς μηχανισμοί εποπτείας, αυτή είναι η γενική δύναμη της εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς καταφέρετε λοιπόν ε, και εποπτεύετε την συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών, όχι μόνο τη διμερή, αλλά και στα πλαίσια του INSENT, αυτού του σκιώδους κοινοτικού θεσμικού οργάνου που επισήμως δεν υπάρχει. Τι άλλο θέλω να ρωτήσω. Α, και μία ακόμη ερώτηση, τελευταία αυτή. Είχαμε εδώ τον εκπρόσωπο της, ε, του, του Βελγικού Φορέα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων στην ε, συνεδρία που είχαμε για την Belgacom και η αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων του Βελγίου φαίνεται ότι είναι πολύ στρατευμένη, πολύ στα πράγματα, μαχητική η υπηρεσία αυτή και εντυπωσιάστηκα γιατί με διαβεβαίωσε εκπρόσωπο αυτής τη υπηρεσία ότι δεν υπήρχε καμία παραβίαση των ε, δεδομένων, ε, κάτι που είναι μάλλον απίθανο, τουλάχιστον αναλυθοφανέ. Μήπως θεωρείτε ότι και αυτή η υπηρεσία προστασία δεδομένων, προσωπικών δεδομένων ε, δεσμεύεται από κάποια ομερτά, από κάποιο απόρριτο, ε, σας έχει επισημάνει μια τέτοια παραβίαση. Αυτά και θα δώσω το λόγο στους Καλεσμένου μας με τη σειρά που έθεσα τις ερωτήσεις, πρώτα στη Δανία και μετά στους Βέλγους συναδέλφου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις ερωτήσει και ευχαριστώ που παίξατε και το ρόλο του δικηγόρου του διαβόλου. Αυτό με διασκέδασε και το απόλαυσε και στην προηγούμενη μα συνεδρίαση. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και πολύ εύστοχες και ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις και πολύ χρήσιμη και για μένα η συνεδρίαση. Ρωτήσατε αν ασκήθηκαν πιέσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Δανία. Δεν το πιστεύω. Εμείς θεωρούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ ισχυρός μας σύμμαχος, έχουμε πολύ στενή συνεργασία και πιστεύω ακράδαντα ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον οι Αμερικανοί να πιέζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις δανεικές αρχές σε ό,τι αφορά την εποπτεία ή δεν αποτρέπουν τις δανεικές αρχές από το να επεκτείνουν αυτή την εποπτεία τους στις μυστικές υπηρεσίες. Και μάλιστα το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί να είναι κατά της συνεργασίας των, με τις υπόλοιπες χώρες ή κατά της εφαρμογής αντίστοιχου συστήματος εποπτείας και από τις σύμμαχες χώρες. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο έχουμε τόσο υψηλό επίπεδο εποπτείας στη Δανία. Αυτό είναι ο πολιτικός συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε, αλλά δεν υπάρχουν και τεκμήρια, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ιδανικές μυστικές υπηρεσίες ή η ιδανική υπηρεσία πληροφοριών κάνουν πράγματα που δεν δικαιούνται. Δεν έγινε και συζήτηση ούτε στη δημοσιογραμμή και δεν ασκείται πίεση στους πολιτικούς. Θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν υπάρχει ισορροπία στο σύστημα και μπορεί να είναι αυτή η προσωπική μου γνώμη, αλλά δεν υπάρχει πίεση για να αλλάξουν οι μηχανισμοί, οι υπηρεσίε εποπτείας ε, στο Κοινοβούλιο ή η ανεξάρτητη υπηρεσία εποπτείας που θεσπίστηκε πέρυσι με το νέο νομοσχέδιο. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να στοιχειοθετούν ε, παράτυπη δράση, κατάχρηση εκ μέρους των δανεικών μυστικών υπηρεσιών ή παράβαση του νόμου εκ μέρους των δανεικών μυστικών υπηρεσιών. Και από τη στιγμή που δεν συγκεντρωθούν τέτοιες αποδείξεις για τα σταλίες της μυστικής υπηρεσίας δεν πρόκειται να ασκηθεί πίεση για την αλλαγή του συστήματος. Φαίνεται ότι τίποτα δεν είναι σαθρό στο βασίλειο της Δανημαρκίας, έτσι. Ο κύριος Δεντέκερ. Ευχαριστώ σε ό,τι αφορά ε, τις υπηρεσίες ε, και το σκάδαλο πρίσμα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία οποιαδήποτε συνενοχή των δικών μας μυστικών υπηρεσιών ή γνώση των δικών μας μυστικών υπηρεσιών και μία ενημέρωση της κυβέρνησης. Και όταν βλέπουμε, όταν βλέπουμε τη, το θυμό, την οργή της α, ε, Γερμανίδας Καγκελαρίου ε, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν την παρακολούθηση και δεν ενημέρωσαν την καγκελάριο. Δεν πιστεύω ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Η συνεργασία τους με τους Αμερικανικές. Τώρα, η NSA είναι στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών του ΝΑΤΟ γνωρίζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Τώρα από εκεί να θεωρήσουμε ότι υπάρχει συνενοχή ή είχαν γνώση της κατάστασης, πολύ αφεβάλλω. Σε εμά βέβαια τώρα ξεκινάει η έρευνα και θα δούμε αν κάποια βελγική υπηρεσία πληροφοριών είχε γνώση της κατάστασης. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι ε, αυτό που συνδέεται κυρίως με αυτή την κατάσταση είναι πρώτα απ' όλα η αφέλεια των ευρωπαϊκών χωρών γιατί η Ήπειρος μας έχει ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμού στον κόσμο εξαιτία του φιλερινικού μας χαρακτήρα. Και μερικές φορές με μεγάλη αφέλεια ε, ε, αντιμετωπίζουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Μερικές φορές οι εθνικές κυβερνήσεις ε, λειτουργούν με βάση τα εθνικά συμφέροντα. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένος ότι μια ωραία πρωία θα διαπιστώσουμε ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες ε, κατασκοπεύουν άλλες ε, ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα όχι σε μικρή κλίμακα αλλά κατά πάσα πιθανότητα σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό θα πρέπει να δούμε κατά μέτωπο. Και εκεί θα πρέπει να διενεργηθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια και αντίστοιχος έλεγχος και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Τώρα, από τη μια λοιπόν είχαμε αυτή την ε, ε, αφέλεια, την αγαθότητα των ευρωπαϊκών χωρών, αφετέρου τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Και ο πειρασμό των μυστικών υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τι προηγμένε τεχνολογίε χωρί κατά να ενημερώνουν και τι κυβερνήσει του. Δεν είμαι 100% σίγουρο ότι οι μυστικές υπηρεσίες, η NSA εξήγησε στον κύριο Ομπάμα κατά λεπτός ε, τις δραστηριότητες της. Πολύ πιθανό να γνώριζε, αλλά πολύ πιθανό και να μην το γνώριζε ο πρόεδρος Ομπάμα. Γι' αυτό είναι και σημαντική εποπτεία από το Αμερικανικό Κογκρέσο των Μυστικών Υπηρεσιών. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχο υπάρχει στι ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά είναι σχετικά κλειστός και ελεγχόμενος για να μπει κανείς στην Επιτροπή Ελέγχου ε, και Εποπτείας των ε, Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών ε, είναι σημαντική πολιτική αναγνώριση και μεγάλο σεβασμός. Ίσως και αυτό το σύστημα στις Ηνωμένες θα πρέπει να εξελιχθεί και ίσως αυτή θα είναι η συνέχεια γιατί δεν φαντάζομαι ότι οι Αμερικανικές αρχές είναι ιδιαίτερα υπερήφανες για τις αποκαλύψεις που έγιναν και χάρη και στον Σνόουδεν, γιατί χάρη στον Σνόουδεν ε, ε, μάθαμε πολύ περισσότερα, θα πρέπει να τα ελέγξουμε και να εξακριβώσουμε την ε, αλήθεια τους, αλλά θα πρέπει να το δούμε και πιστεύω ότι και στο ΝΑΤΟ θα γίνει μια τέτοια ζήτηση μεταξύ των συμμάχων, γιατί ούτε και εγώ θέλω να φανώ αγαθός και αφελής. Ο κύριος Ραπάγη. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος ε, Δεντέκερ. Οι έρευνές μας τώρα συνεχίζονται και θα δούμε την επόμενη εβδομάδα και στο μέλλον ποια θα είναι τα πορίσματά τους. Τώρα, ρωτήσατε τι γνώριζαν οι μυστικές υπηρεσίες. αν όφυλα να γνωρίζουν την κατάσταση. Και αν έκαναν μια ανάλυση του κινδύνου, δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας τους μετά τις υποθέσεις SWIFT και Shellon. Μήπως θα όφυλαν ή θα δίναντο οι μυστικές υπηρεσίες να σκεφτούν ότι με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις θα υπήρχε και περισσότερες δυνατότητες. Αυτό το ερώτημα καλούμαστε να απαντήσουμε, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει στην απάντηση. Άλλωστε δεν έχουμε ενδείξεις που να μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι βελικές μυστικές υπηρεσίες με τα μέσα που έχουν μπορούν να παρακολουθούν την κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, εκτό ε, μικροφώνου δυστυχώ στο σχόλιο τη κυρία Σίνβελτ, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ε, πληροφοριών, αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο. Έχουμε συνεργασία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών. Ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τις στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες που αυτές έχουν επαφή με το ΝΑΤΟ. Ενώ οι πολιτικές μυστικές υπηρεσίες ε, περιορίζονται την κατάσταση στο Βέλγιο και ενεργοποιούνται στη βελγική επικράτεια. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ακόμη τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Πάντως, αν θέλουμε μία απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει κατακλείδη στην παρουσίασή μου. Θα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες και στα Εθνικά Κοινοβούλια, ώστε να θεσπιστούν αποτελεσματικοί κοινοβουλευτικοί μηχανισμοί εποπτείας. Και να μην έχουμε απλώ υπηρεσίε που δεν έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που θα πρέπει να παίρνουν από τι κυβερνήσει για να λαμβάνουν τι πληροφορίε. Όλε αυτέ οι προσπάθειε θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, Επιτροπή για την Προστασία της Ιδιωτικής Σφαίρας, ε, είχατε εκπρόσωπό της ε, στην ε, συνεδρίασή σας. Δεν ξέρω τι πληροφορίες σας έδωσαν. Εμείς έχουμε κάποιες επαφές μαζί τους, αλλά κυρίως η Επιτροπή αυτή ασχολείται με την προστασία της προσωπικής ζωής. Δεν ξέρω τώρα αν έγινε ε, κατάχρηση τέτοιων προσωπικών δεδομένων ερήμην των υπηρεσιών. Μερικά στοιχεία μας διαφεύγουν. Πάντως έχουμε και δικαστικές έρευνες που εκτιλήσονται και θα δούμε τι θα γίνει και στην υπόθεση Belgacom και σε άλλες υποθέσεις. Γιατί είχαμε καταγγελία και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τον Πρωθυπουργό για παγίδευση και παραβίαση και των δικών τους ε, επικοινωνιών. Δεν ξέρουμε από ποιον και γιατί, αλλά εκτελήσετε για το θέμα αυτό δικαστική έρευνα. Ευχαριστώ. Περνάμε στις ε, τελευταίες ερωτήσει που θα ακούσουμε σήμερα για να Αλμπρέχτη. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω τον καλό ή τον κακό μπάτσο. θα σας μιλήσω ως συνάδελφο. Χαίρομαι που είστε εδώ. Και χαίρομαι που αναφέρατε την διακήρυξη των Βρυξελών και για το ότι ζητάτε κοινή δράση. Αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Από αυτήν εδώ τη συνεδρίαση και από την έκθεσή μας ελπίζω που θα είναι έτοιμη αρχές ε, του επόμενου έτους αλλά πρέπει να πω επίσης κοιτώντας ε, την κατάσταση ε, υπάρχει η συνθήκη και έχουμε γραπτές απαντήσεις από τις δικές σας και τις δικές μας κυβερνήσεις που λένε πως δεν θα καταθέσουν εδώ πέρα. Η εθνική ασφάλεια είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω το εξής. Κύριε Λεόνσεν, ξέρετε τι είναι. Ίνσεν ασχολείστε με τη συνεργασία μυστικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασχολείστε με τα θέματα του ποιοι κανόνες εφαρμόζονται γιατί πρέπει να σου πω έψαξα για νομική βάση για αυτή τη συνεργασία και δεν υπάρχει νομική βάση είναι και παραβίαση των συνθήκων σύμφωνα με την ερμηνεία των κρατών μελών δηλαδή χωρίς τη δική σας τη βοήθεια δεν θα γίνει τίποτα και με συγχωρείτε κιόλας αλλά είναι σημαντικό γιατί πολιτικά τα επόμενα χρόνια πρέπει να γίνει κάτι γιατί ο κόσμος ρωτάει εμάς τους βουλευτές, ευρωβουλευτές και βουλευτές. Οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάνω από τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις. Δεν τους αγγίζει κανείς. Δεν αναπορεί κανείς ε, το ότι ψηφίζει ο κόσμος λαϊκιστές που τους λένε πως ε, όλα αυτά είναι μπουρδες. Για τη Δανία, να επισημάνω. Πως εδώ στην πρώτη μας ακρόαση είχαμε τον Ντάνκεβ Κέμπελ, δημοσιογράφο, ο οποίος μας είπε σε σχέση με τα έγγραφα Σνόντον που δεν έχει αμφισβητήσει κανείς πως η Δανία έχει πρόγραμμα συνεργασίας με την ΕΝΕΣΕ ονόματι Δυναμό το οποίο εξετάζει, κοιτάει το, το, τα υποθαλάσσια καλώδια, με κάποιο τρόπο τα παρακολουθεί και ε, παρακολουθεί όλες τις πληροφορίες γενικώς, αδιακρίτως. Αυτό είναι παραβίαση δεν ξέρω, του διεθνούς δικαίου, του εθνικού, του οπωσδήποτε της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του άρθρου 10 της ε, Συνθήκης ε, και της ε, νομολογίας του δικαστηρίου που είναι θεμέλια, θεμελιώδης αρχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Και επίσης, μην ξεχνάμε, και την συνεργασία που είναι επίσης θεμελιώδης ε, αρχή σύμφωνα με τον νόμο. Δηλαδή, η συνεργασία αυτή είναι τελείως αντίθετη με τις διμερείς συμφωνίες που αναφέρατε και δεν βλέπω πραγματικά πως οι επιθέσεις ε, ε, Βρετανών, Βρετανικών αρχών όπως η επίθεση αυτή σε, υποδομών, σε υποδομές άλλων κρατών μελών, όπως ο σερβερ του Facebook στη Σουηδία ή η επίθεση σε εταιρείε άλλων κρατών. Πώς είναι δυνατόν να γίνονται, πρέπει να κινητοποιηθούμε εδώ πέρα και θα ήθελα πραγματικά να ξέρω τι κάνουμε, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ζητάμε να μην γίνει τίποτα άλλο. Ε, Αλλιώς ε, τι θα εφαρμοστεί η διακήρυξη των Βρυξελών ε, από τις κυβερνήσεις μας. ποιο είναι το επόμενο βήμα. Απλά βγάζουμε μια διακήρυξη και λέμε ναι εντάξει κάνουμε κάτι αλλά στην πράξη τίποτα. Επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε το τι είναι η, η, η ξένη αυτή ασφάλεια όπως αναφέρθηκε. Ε, η γερμανική αρμόδια υπηρεσία θεωρούσε το ίντερνετ ως εξωτερικό, εκτός γερμανικής επικράτειας. Αν το κάνει αυτό η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών, σημαίνει πως φοβούνται πραγματικά την κατακραυγή, έτσι. Πρέπει να αρχίσετε λοιπόν κάποια έρευνα και στις ε, χώρες σας. Και θα ήθελα να μάθω αν ε, ισχύει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ναι, Κοιτάξτε, σκέφτομαι πως πάρα πολλοί λένε ε, δεν πρέπει να δώσουμε άλλες αρμοδιότητες στις Βρυξέλλες γιατί γίνονται υπερκράτος. Αλλού είναι το υπερκράτος όμως. Κύριε Λάριτσεν, Ντεντέκερ, σας ακούμε. Κύριος Λάριτσεν. Ένας από τους προηγούμενους ομιλητές ε, είπε πολλές φορές ουδέν σχόλιον. Το ίδιο θα αναγκαστώ να πω και εγώ σε κάποιες ερωτήσεις για το θέμα του δυναμό ας πούμε και τη συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. δεν μπορώ να σχολιάσω. Και να ήξερα δεν θα μπορούσα να σας πω έτσι. Για την Ίνσεντ δεν ε, υφίσταται τέτοια συζήτηση στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Ίσως θα έπρεπε να το συζητάμε το θέμα. Και τα δύο θέματα αυτά, αλλά όπως είπα δεν το συζητάμε. Επίσης και το κοινοβούλιο μας είναι διχασμένο για το εάν πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτική εποπτεία. Κάποιοι λένε πως εάν κάνουμε κάτι τέτοιο είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Ίσως καλύτερα είναι ο υπουργό μόνο να ξέρει. Και οπωσδήποτε ο υπουργό γνωρίζει. Ε, αυτό σας το λέω 110% σίγουρος. Το τι κάνουν οι μυστικές μας υπηρεσίες και τι συνεργασία έχουν με άλλες χώρες κτλ. Και μπορεί να ενημερωθεί. Το σημαίνει όμως πως ε, είναι και υπεύθυνο και κάποιοι ε, βουλευτές λένε πως ε, η καλύτερη λύση είναι ο υπουργός που ξέρει τα πάντα να είναι και υπεύθυνο. Γιατί αν τα ξέρει και η Επιτροπή Υποπτείας, εμέσως γίνεται επίσης συνυπεύθυνη. προβλέπω τον Μπόργκεν, το σύριαλ το αστυνομικό να γυρίσει άλλη, άλλη μια σεζόν με αυτά που λέτε. Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο σύριαλ. Ε, είναι σύριαλ όμως έτσι, δεν είναι η πραγματικότητα. πολύ καλό. πολλοί Σκανδιναβοί βουλευτές έρχονται στην Δανία και λένε θέλουμε να πάμε στο, στο κοινοβούλιο της Δανίας ε, εκεί όπου συμβαίνουν αυτά που δείχνει τον Μπόργεν αλλά και εμείς ε, ένα βαρετό κοινοβούλιο είμαστε στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το θέμα της συνεργασίας. Οπωσδήποτε θα εξτάσουμε την έκθεσή σας. Και θα δούμε και τις ε, συστάσεις σας. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει περιθώριο κάποιας ε, συνεργασίας με τις μεγάλες εταιρείες, Facebook, Google, γιατί οπωσδήποτε δεν ε, ενδιαφέρονται. Δεν έχουν κανένα συμφέρον οι μυστικές υπηρεσίες οποιασδήποτε χώρας να παίρνουν τις πληροφορίες τους. Οπότε και εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε κάτι, να συνεργαστούμε με τις χώρες αυτές. Ε, μιλάμε για στατιστικά, ας πούμε, πόσες φορές οι μυστικές υπηρεσίες, οι αρχές τους ζητάνε να δώσουν στοιχεία. Παραδείγματος χάρη. Οπότε μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα που σας είπα. Σας ευχαριστώ. Σιγά σιγά. Πλησιάζουμε στο τέλος. Κύριε Ντεντέκερ. Σας ευχαριστώ. Ζούμε σε έναν κόσμο που αδιαμφισβήτητα είναι επικίνδυνος και που βλέπει να εξελίσσονται και οι απειλέ. Πριν από 10 χρόνια κανένα δεν μιλούσε για κυβερνοεπιθέσει. Τώρα αποτελούν ε, την. ε, ε του φόβητρο των κυβερνήσεών μας, για τις κυβερνήσεις μας μάλλον, και όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Κίνα και άλλες χώρες που έχουν ε, ε, καταγγελθεί Όλα αυτά τα αποδεικνύουν τα γεγονότα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς οι Ευρωπαίοι, αν συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα άμυνας και ασφάλειας μόνο σε εθνικό επίπεδο, και δεν εξελιχθούμε προς μια πραγματική ευρωπαϊκή άμυνα, θα αποδυναμωθούμε όλο ένα και περισσότερο. Υπάρχουν ε, χώρες ε, όπως η Γαλλία και η Βρετανία που πιστεύουν και που ονειρεύονται ότι εξακολουθούν να είναι υπερδυνάμεις και πάνω σε αυτές τις απειλές δεν είναι πλέον καθόλου. Οι ίδιες όμως θέλουν και επιμένουν να ρυθμίζουν αυτά τα θέματα σε στηρά εθνικό επίπεδο. Και θα ήθελα να σας πω ότι εγώ 25 χρόνια ήμουνα στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και πρόεδρος της Επιτροπής Αμήνης αυτής. Πάει η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, έκλεισε, οι αρμοδιότητες της διαβιβάστηκαν στην Ένωση. Συνέπεια αυτό είναι ότι οι εθνικοί βουλευτές που συμμετείχαν σε μεγάλο αριθμό στο Κοινοβούλιο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αρκετά καλά ενημερωμένοι για τα θέματα αμήνης και ασφάλειας. Και οι υπουργοί έρχονταν σταδιακά στην Σύνοδο στο Παρίσι για να τα εξηγούν όλα αυτά. Τώρα όμως η αρμοδιότητα είναι στην Ένωση και το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά δεν έχει υπάρξει ολοκλήρωση υπάρχει αρμοδιότητα της Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου. Και το, και το Ευρωκοινοβούλιο και οι εθνικοί βουλευτές των Επιτροπών Αμήνης συνεδριάζουν δύο φορές ετησίως. Η κυρία Άστον έρχεται και μιλά 10 και ο κύριος Ράσμουσεν επίσης. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον έλεγχο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα. Είμαστε απείρως λιγότερο ενήμεροι για το τι τρέχει. Και η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, ε, αντί να προοδεύει. Ενώ αντίθετα θα έπρεπε να προχωρήσουμε γρήγορα προς ολοκλήρωση των όσων θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν την ολοκλήρωση της αμυντικής πολιτικής και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρε θα μπορούσαν ήδη να το κάνουν αυτό. Και τα λοιπά, πολύ απεσιόδοξα χρωματίσαμε το ρόλο των μυστικών υπηρεσιών και ότι δηλαδή είναι πάνω από τις κυβερνήσεις. Όχι, βεβαίως και όχι. Καλύτερα είναι να ελέγχονται από την κυβέρνηση και από το κοινοβούλιο, πάντως σίγουρα δίνουν λογαριασμό στην κυβέρνησή τους παντού, γιατί τα ατυχήματα σε αυτούς τους τομείς μπορεί να κοστίσουν πολύ ακριβά στις κυβερνήσεις. Και οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες λοιπόν ε, πληροφόρησης, πληροφοριών μάλλον, το συνειδητοποιούν πολύ καλά και είναι διαρκώ σε επαφή. Μιλάω για τις πολιτικές υπηρεσίες. Οι στρατιωτικές στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και αυτές τα λένε μεταξύ τους. Εσείς καταγγέλλετε την υπόθεση των υποθαλασσίων καλωδίων. Το ανακαλύψαμε αυτό την ε, καιρό του ΕΣΕΛΟΝ. Υπήρξε συμφωνία ανάμεσα είπα και Ηνωμένο Βασίλειο για να παρακολουθούν τα σοβιετικά υποβρύχια ε, που διέστησαν τον Ατλαντικό και με την ίδια αρχή παρακολούθησαν και τα υποθελάσια καλώδια και τους δορυφόρους μετά και το πρίσμ ΝΑΤΟ. Ε, τα ίδια είναι αυτά, δεν είναι κάτι το νέο. Αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα όνειρα υπερβολικής ε, ε, κυριαρχίας, κυρίως από πλευράς των μεγάλων παλιών ετών, είναι εις βάρος της ε, γενικής μας ασφάλειας. Γιατί αυτό που γίνεται εδώ και οι κυβερνοεπιθέσεις και οι παρακολουθήσεις ε, πληροφοριών και, τα, και συνδιαλέξεων κτλ. Εάν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε εθνικό επίπεδο και εμείς οι ίδιοι πέφτουμε θύματα των συστημάτων παρακολούθησης μιας γειτονική χώρας της Ένωσης, αυτό δεν μπορεί παρά να αποδυναμώνει την ευρωπαϊκή συνείδηση των κρατών χωρών, μελών. Αν αρχίσουμε ένας να υποψιάζεται τον άλλον, είναι εξαιρετικά ζημιοκόνο για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη μέσω αυτού του φαινομένου της ολοκλήρωσης για να εξασφαλιστεί η συνέχιση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και να μην πάμε προς την σταδιακή της διάλυση μετά από σοκ και φαινόμενα κρίξεων και κυβερνήσεων που ξαφνικά θα σοκαριστούν ε, ε, και θα ε, λειτουργήσουν επιθετικά εις βάρος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ραπάγια, έχετε να προσθέσετε κάτι στο τελευταίο μας ομιλητή. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπε ο κύριος Δεντέκερ. Ίσως θα μπορούσατε να απαντήσετε σε μία συγκεκριμένη ερώτηση για να ολοκληρώσουμε τι θα γίνει μετά τη διακήρυξη των Βρυξελών, ποια θα ήταν η συνέχεια που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Συμμετείχα στην ε, ίδρυση αυτού του φόρουμ, που είναι ένα φόρουμ κοινοβουλευτικού ελέγχου των ε, μυστικών υπηρεσιών. Και χαίρομαι που κάθε χρόνο περνάει όλο και περισσότερες χώρες ε, προσχωρούν στο φόρουμ αυτό. Και φαίνεται ότι Αργά αλλά σταθερά σημειώνουμε πρόοδο. Και μετά τις τελευταίες εξελίξεις πιστεύω ότι τα κοινοβούλια που έχουν τέτοια δυνατότητα ελέγχου θα καταλήξουν σε κοινέ πρωτοβουλίες που θα αναδειχθούν στις επόμενες συνεδριάσεις του φόρουμ αυτού. Γιατί σε κάθε συνεδρίαση, σε κάθε διάσκεψη ήμασταν όλο και πιο ευτυχείς. Κάθε φορά είχαμε μία ποιοτική αναβάθμιση και μία πρόοδο. Αλλά έχουμε ακόμη φυσικά πολύ δρόμο μπροστά μας. Και μάλιστα η έκθεση και της δικής της επιτροπής σου θα είναι χρήσιμη και θα έχει απήχηση και στο φόρουμ αυτό. Θα μπορούσα να προσθέσω εδώ, γιατί αναφερθήκατε πολλά και στη συνεδρίαση και διακήρυξη των Βρυξελών του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2010 αλλά είχαμε και στη Βόνη τον Οκτώβριο του 2011 συνεδρίαση και το 2012 και 2013 δεν έγινε καμία τέτοια διάσκεψη. Αυτό που θα μπορούσατε λοιπόν να κάνετε εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να δώσετε νέα όθηση στη διαδικασία, να γίνει μια επανέναρξη της διαδικασίας, ώστε να έχουμε και πάλι συνάντηση αυτών των ελεκτικών οργάνων, γιατί ο κύριος Δεντέκερ αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί. Εγώ συμμετείχα σε ορισμένες από τις ε, διασκέψεις, ε, όχι σε όλες. Φαίνεται ότι με το πέρασμα του χρόνου ενισχυόταν η εμπιστοσύνη και μάλιστα στη διάσκεψη της Βόνης για πρώτη φορά οι βουλευτές συζήτησαν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τους κανόνες που θα πρέπει να θεσπίσουμε ώστε να θέσουμε ένα τέρμα στον κανόνα της ε, τρίτης υπηρεσίας. Μήπως θα πρέπει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να ακυρώσουμε αυτόν τον κανόνα ώστε να μην μπορεί να τον επικαλείται η μυστική υπηρεσία, μια μυστική υπηρεσία. Νομίζω ότι είναι χρήσιμος αυτός ο κανόνας, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται με μέτρο και υποπεριορισμό. Και από αυτήν την άποψη θεωρώ ότι η Επιτροπή σας θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να ξαναθέσει σε, στις ράγες αυτή τη διαδικασία. Γιατί άλλο η συνεργασία σε διμερές επίπεδο μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών και άλλο ο έλεγχος που θα πρέπει να ασκείται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και να εκπορεύεται είτε από τα εθνικά κοινοβούλια είτε από το ευρωπαϊκό. Αυτά. Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση, εκτός και αν ε, επήγεστε να κάνετε και μια τελική δήλωση. Αυτές οι απογευματινές ε, συνεδρίες πέμπτης ε, είναι πολύ δύσκολες και για τους βουλευτές και για το προσωπικό, γιατί έχουν όλοι πτήσεις να προλάβουν. Από άψη και οργάνωση είναι πολύ δύσκολες αυτές οι συνεδριάσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά και πάλι να εκφράσω μία απογοήτευση με, με απογοήτευσε ο, ο Δανός συνάδελφος, γιατί εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούσαμε ότι αυτή η σειρά το Μπόργεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Όχι, ο Πρωθυπουργό είναι πραγματικός. Το σύριαλ είναι φανταστικό. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Ραντεβού και πάλι για τη συνέχεια τη Δευτέρα το απόγευμα στο Στρασβούργο.